Okay. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στην τακτική μας συνεδρίαση. Στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης, την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό Λίδια Μούζ που είναι υπουργό ε, Υγεία του Λουξεμβούργου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητές σας και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών για τις προτεραιότητές σας αλλά και τις προοπτικές κάποιων θεμάτων που βρίσκονται επιτάπητος εδώ και πολύ καιρό και θέλουμε επιτέλους να τα διεκπαιρεώσουμε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Υπουργό Μούτς για να μας κάνει την εισαγωγική της ομιλία και μετά θα έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων. Το πρώτο με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και το δεύτερο με τους λοιπούς ευρωβουλευτές. Κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με τιμά ιδιαίτερη η παρουσία μου εδώ. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, γνωρίζετε ότι μια Προεδρία δημιουργεί ανέκαθεν μια μείζωνα πρόκληση για ένα κράτος μέλος, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και μια καταπληκτική ευκαιρία ε, για συμμετοχή στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της. Είναι αλήθεια ότι το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει για 12η φορά τα ενία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτή η Προεδρία λαμβάνει η προεδρια λαμβανει χωρα σε ιδιαίτερες συνθήκες γιατί έχουμε μια Ευρώπη που ακόμη πασχίζει να εξέλθει από την κρίση, να ανακάμψει και ταυτόχρονα μια Ευρώπη με γυράσκοντα πληθυσμό κάτι που δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στη δημόσια υγεία. Επίσης έχουμε μια Ευρώπη με ένα νέο Κοινοβούλιο που μπήκε πια κανονικά στο ρυθμό του και έχουμε και μία νέα επιτροπή που στηρίζει τις δράσεις της ε, σε μία νέα μέθοδο εργασίας και μία προσέγγιση που στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον και ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές αλλά και από καινοτομίες. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό η δημόσια υγεία, το θέμα της δημόσιας υγείας και ο ίδιος ο ασθενής να μην ε, παραγωνιστούν από τις προτεραιότητές μας. Και για αυτό το λόγο η, Πορτογαλ... η Λουξεμβουριανή Προεδρία έθεσε τις εργασίες της στον αστερισμό του ασθενούς και της καινοτομίας. Πρόκειται για μία ποδό που συνάδει πλήρως και με το γενικό θέμα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας που είναι μία ένωση για τον πολίτη. Γι' αυτό ακριβώς υιοθετήσαμε μία προσέγγιση που θέτει τον ασθενή στο επίκεντρο των συζητήσεων. και αυτό το θέμα επαναλαμβάνεται σε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Σήμερα το πρωί με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο τομέα της δημόσιας υγείας, των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αλλά και στο θέμα της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων. Ξεκινώ λοιπόν από την δημόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της δημόσιας υγείας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ένα ζήτημα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Το θέμα της εξατομικευμένης ιατρικής. Πρόκειται για ένα θέμα που συνδυάζει θαυμάσια τον ασθενή με την καινοτομία. Η εξατομικευμένη ιατρική ξεκινά από τον ασθενή θα πρέπει όμως ε, να εξασφαλίσουμε και ισότιμη πρόσβαση σε τέτοιου είδους ε, καινοτόμες θεραπείες που κατά τη γνώμη μου θα δημιουργήσουν την επανάσταση και θα μεταρρυθμίσουν ρηξικέλαστα την ιατρική μας. Η εξατομικευμένη ιατρική έχει ένα τεράστιο δυναμικό για να βελτιώσει την υγεία των ασθενών με πιο στοχευμένες θεραπευτικές αγωγές που θα μειώσουν αισθητά τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Ταυτόχρονα η ιατρική αυτή θα εξασφαλίσει παράταση μιας ποιοτική ζωής στον ασθενή. Επίσης θα συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά συστήματα υγείας. Στις 8 Ιουλίου, πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, έλαβε χώρα μία διάσκεψη υψηλού επίπεδου στο Λουξεμβούργο με θέμα την πρόσβαση των ασθενών στην εξατομικευμένη ιατρική και στην διάσκεψη αυτή δόθηκαν κάποιες απαντήσεις στις πολυάριθμες προκλήσεις που ανακύπτουν και που εμποδίζουν ε, μέχρι στιγμής την ε, ένταξη των καινοτόμων θεραπείων στην κλινική πράξη. Κάτι που κατά τη γνώμη μου αποτελεί εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στα ωφέλη της προσωποποιημένης, της εξατομικευμένης ιατρικής. Τα βασικά μηνύματα της ε, διάσκεψης αυτής θα αποτελέσουν τη βάση των συμπερασμάτων που θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας ε, στις 8 Δεκεμβρίου. Μια άλλη προτεραιότητα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας θα είναι η άνοια. Ένα τομέας που θέλουμε να εξεταστεί υπό το φως ε, καινοτόμων ε, προσεγγίσεων και προς όφελος των ε, πασχόντων ε, από άνοια. Βρισκόμαστε σε μια γυράσκουσα Ευρώπη και ο αριθμός των ασθενών, των πασχόντων από άνοια αυξάνει σταθερά. Όχι μόνο από άνοια αλλά από και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Αυτές οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες βρίσκονται σε αναδική πορεια πορεία δυστυχώς, δημιουργώντας ένα πραγματικό κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα. Η Προεδρία μας θα εγκύψει το θέμα της άνοιας και θα την αναλύσει ως κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο που χρήζει πολυτομεακής απάντησης. Θα ήθελα λοιπόν να εξετάσω τον χρήσιμο ρόλο που έχει η δευτερογενής πρόληψη και η μεταδιαγνωστική στήριξη για να μειωθεί η επιβάρυνση ε, της φροντίδας των πασχόντων από Επίσης θέλω να εξετάσω την προστιθέμενη αξία που θα έχει μία κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ε, κοινή αξιοποίηση και την ανταλλαγή των ε, καλών πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται σε πολλά κράτη-μέλη. Τα σχετικά συμπεράσματα επίσης ε, θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας του Δεκεμβρίου. Η Προεδρία μας θα κάνει επίσης και έναν απολογισμό της εφαρμογής της οδηγίας για την διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη με βάση την έκθεση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται ο νούπο, ελπίζω πριν τις θερινές διακοπές. Και σήμερα, δύο χρόνια μετά την εκπνοή της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας, είναι και καινή ώρα να καταρτήσουμε ένα πρώτο απολογισμό της εφαρμογής της οδηγίας και αν είχε, να δούμε αν είχε ένα θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό κινητικότητας και αν όντως επέτρεψε στους ασθενείς να βελτιώσουν την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή να διαπιστώσουμε τι συνέπεια είχε η οδηγία στο διοικητικό φόρτο και για τους ασθενείς και για τις ε, εθνικές αρχές και πώς χειρίστηκαν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη νέα οδηγία. Επίσης, ε, το σκέλος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ιδιαίτερα μεταξύ όμορων χωρών. Όλα αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία του απολογισμού της εφαρμογής της οδηγίας για την διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη. Επίσης, ε, θα συνεχίσουμε ένα θέμα που ήταν σημαντική προτεραιότητα της Λετωνικής Προεδρίας και πολύ σωστά και εννοώ τη μείωση των ε, βλαβών που οφείλονται στην κατάχρηση του αλκοόλ. Οι Υπουργοί έστειλαν μια ηχηρή έκκληση και σχεδόν ομόφωνη έκκληση στο άτυπο συμβούλιο στη Ρήγα που έγινε τον Απρίλιο και το ηχηρό αυτό μήνυμα έλεγε ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για το αλκοόλ. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ελήφθη το μήνυμα που εστάλει στη Λοξεβουριανή Προεδρία και το σχέδιο των συμπερασμάτων μας ήδη συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις αρχές Ιουλίου. Τα συμπεράσματα αυτά καλούν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις εθνικές προσπάθειες για να περιορίσουν τις βλάβες εξαιτίας της κατάχρησης του αλκοόλ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναπτύξει για το 2016 μία ειδική στρατηγική για το αλκοόλ. Και περιμένουμε από τον Επιτρόπο Ανδριουκάητης να δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την έκκληση με χειροπιαστές δράσεις που περιμένουν τα κράτη-μέλη. Φυσικά περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδοκαιτοθεσία σε ό,τι το θρεπτικό περιεχόμενο των ενοπνευματοδών ποτών. Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του 2011 για την ενημέρωση των καταναλωτών ε, για τα τρόφιμα. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα αποτελέσει την ευκαιρία για τον απολογισμό μας ως προς τα διδάγματα που αντλήσαμε από τη διαχείριση της, επιθυμίας, της επιδημίας έμπολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαζί με τον Πίτρο Ανδριουκάητης θα καλέσω τους Υπουργούς Υγείας σε μια υπουργική διάσκεψη στην οποία θα καλέσουμε και αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η διάσκεψη αυτή θα δώσει έμφαση στις υγειονομικές πτυχές της επιδημίας. Θέλουμε να εντοπίσουμε τα διδάγματα που είναι απαραίτητο για να ενισχύσουμε την υγειονομική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση μελλοντική επιδημία. Και οι πρόσφατε εξελίξει στη Λιβυρία κατέδειξαν ότι δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο ιό έμπολα και υπάρχει ο κίνδυνος για να ξεσπάσει μια νέα επιδημία. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε θέση και να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα που θα υιοθετήσουμε στο Συμβούλιο της 8ης Σεπτεμβρίου. Θα περάσω τώρα στα φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές. Έχουμε καταρχήν τη μεταρρύθμιση σε σχέση με τον ιατρικό εξοπλισμό. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει τα μάλα και για μας ως Προεδρία είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και φυσικά θα αποδώσουμε στο θέμα αυτό μια ιδιαίτερη και σημαντική προσοχή. Είναι μια κέρια και κρίσιμη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε για το θέμα αυτό. Στις 28 Ιουνίου έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τις ρυθμίσεις για αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Πρέπει λοιπόν να ε, αντιμετωπίσουμε τις ε, αιτιολογικές ε, σκέψεις που βρίσκονται στο, στην πρότασή μας για να ξεπεράσουμε κάποιες συνέχειες ίσως σε ό,τι αφορά τη διατύπωση γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν διατυπωθεί και έχουν τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Θα περάσουμε μετά στον τριγωνικό διάλογο με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, το ταχύτερο δυνατό και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να ακολουθήσουμε τις απαραίτητες ε, γενικές ε, ρυθμίσεις. Με τις επαφές μου στο με το Κοινοβούλιο έχω κατανοήσει ότι ακολουθούμε τις ίδιες κατευθύνσεις. Θέλουμε να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να είναι σαφές και, τα, και να επιτρέψει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, συγχρόνως ενθαρρύνοντας μια αγορά η οποία θα είναι καινοτόμα στα θέματα αυτά. Επίσης, έχουμε τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα, πιστεύω θα έχετε ένα σημαντικό το ταχύτερο θα μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν μία λύση με την νομοθετική διαδικασία και έτσι να προετοιμάσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη αδημονία να δούμε τι θα προκύψει από όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα την υγειονομική ασφάλεια και την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα αυτό. Περιμένουμε να υπάρξουν και περισσότερες ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά, ξεκινώντας από την κλωνοποίηση και τις τεχνικές ζωικής αναπαραγωγής. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι σε εξέταση από το Συμβούλιο και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέγονται από το Συμβούλιο. Όλα αυτά αποτελούν ένα πακέτο το οποίο είναι αδιάσπαστου χαρακτήρα. Και πιστεύουμε ότι η έγκριση αυτών των τροπολογιών θα είναι ένα σημαντικό ατού για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και την περαιτέρω εξέλιξη σε αυτό το φάκελο. Με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να παραπέμψουμε αυτά τα θέματα στις υπηρεσίες του Συμβουλίου, αλλά φυσικά εξαρτώμεθα από τις εργασίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ένδυση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η δυνατότητα η οποία προσφέρεται αυτό το κείμενο, αυτό το οποίο παρουσιάζεται για τα κρατημέλη, είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν και πλήρως την εφαρμογή στο έδαφος τους της χρήσης <clears throat> γενικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Λοιπόν και η Κομισιόν μέσα στις επιλογές που έχουν γίνει δίνει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να έχει ένα αποφασιστικό ρόλο για τα θέματα αυτά και για την κατεύθυνση που θα αναλάβουν αυτές οι εργασίε. Έχουμε καταγράψει επίσης τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από το Συμβούλιο για τα Αγροτικά Θέματα την προηγούμενη Δευτέρα σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος αντικτύπου και καλύτερη διευκρίνηση ορισμένων νομικών πλευρών για τα πρακτέα κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουργιακής Προεδρίας θα δώσουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον στην παρακολούθηση των συζητήσεων στις διάφο στους διάφορους φορείς του Κοινοβουλίου. Η έγκριση των νέων τροφίμων, τη λεγόμενη οδηγία Novel Food. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα ως Λουξεμβουργική Προεδρία Στις 25 Ιουνίου υπήρξε μια ψηφοφορία κατά στην Επιτροπή σας, την οποία χαιρετίζει η Προεδρία και φυσικά κατανοούμε τα θετικά στοιχεία της πρότασης αυτής. Είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία έγκρισης των λεγόμενων νεοφανών τροφίμων. Η ψηφοφορία αυτού του Κοινοβουλίου κατέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης, το οποίο θα επιτρέψει <clears throat> να δημιουργήσουμε ένα εξυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για τα νέα τρόφιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και αν το κείμενο αυτό εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι μπορεί το ταχύτερο να εγγραφεί στην ημέρηση διάταξη του Συμβουλίου για οριστική έγκριση. <clears throat> Έρχομαι τώρα στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και εδώ η Λετωνική Προεδρία έχει καταφέρει να κάνει σημαντικές προόδους για την πρόταση αυτή και εδώ περιλαμβάνει αυτή η πρόοδος και μερικά σημεία τα οποία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα και για εσάς αλλά με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εστιάσουμε καλύτερα την προσοχή μας στα διάφορα σημεία τα οποία παραμένουν ακόμα εκκρεμή παραδείγματο χάρη τον ρόλο και της υπευθυνότητα του επίσημου κτηνιάτρου. Προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια εντολή σε επίπεδο κορεπέρ το δυνατό για να ξεκινήσουμε τη συζητήση με το Κοινοβούλιο ή δυνατόν και αν θέλει ο Θεός από τον Σεπτέμβριο. Στόχο είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία, μια ταχεία συμφωνία Δευτέρας Ανάγνωσης. Αυτή είναι και η ελπίδα μας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι διαπραγματεύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα θα είναι επικοδομητικές και καρποφόρες. Και είμαστε φυσικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και έχουμε το τέλος στο θέμα της ετικετοθεσίας στα τρόφιμα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες για το θέμα αυτό από το 2008 και φυσικά καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια έχουν περάσει. Ο κανονισμός 1169-2011 εφαρμόζεται ήδη και είναι ορατά τα αποτελέσματά του. Για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που έχουν ήδη νέες ετικέτες οι οποίες είναι πιο αναγνώσιμες και πιο πλήρες σε πληροφοριακό επίπεδο στα πλαίσια αυτά η Κομισιόν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα, δώσει, θα περατώσει τις εργασίες σε σχέση με την έκθεσή του για την ε, έκθεση που αφορά την παρουσία λιπαρών οξέων σε ορισμένα τρόφιμα που θα έπρεπε ήδη να είχε δημοσιευτεί το Δεκέμβριο του 2014. Επομένως, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί στο άτυπο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο με στόχο να σφιγμομετρηθούν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο ώστε να υπάρξει η απαραίτητη προστασία των καταναλωτών για να γνωρίσουν την παρουσία αυτών των λιπαρών οξέ, οξέων στα τρόφιμα αυτά. Είτε μέσω της ετικετοθεσίας, είτε μέσω της ε, ρύθμισης για ανώτατα όρια παρουσίας των ε, λιπαρών οξέων, είτε μέσω εθελοντικών μέτρων. Τα μη και κορεσμένα λοιπόν λίπαρα οξέα θα αντιμετωπιστούν και μέσα στην ανταλλαγή απόψεων του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ στις 8 Δεκεμβρίου και η συζήτηση αυτή ελπίζω θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να αποφασίσουν καταρχήν σε σχέση με το πλαίσιο το ρυθμιστικό πρέπει να διέπει αυτά τα μη διακορεσμένα λιπαρά οξέα. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγεία των πολιτών μας. Για να κλείσω. Θα ήθελα να σας ε, διαβεβαίωσω κυρίε και κύριοι ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είσαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών και επομένως εναπόκειται σε εσά να αρθρώσετε το σύνολο των ερωτημάτων που ενδιαφέρουν τους πολίτες μας κατά διάρκεια των επόμενων έξι μηνών λοιπόν θα κάνω ό,τι πεθάει από το χέρι μου τα χέρια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινό όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και έτοιμοι είμαι να απαντήσω σε όλα τα θέματα τα οποία τυχόν θέλετε θέση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you very much for your introductory statement Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, καθώς και για τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας σας για το επόμενο εξάμεινο. Θα ξεκινήσουμε άμεσα το πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους εκπροσώπους των ομάδων και ξεκινάμε τον Πίτερ Λίζε εξ ονόματος του ΕΛΟΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου για την παρουσίασή σας και για τη δέσμευση που έχετε καταδείξει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την νομοθεσία στον τομέα αυτό και για αυτά που μπορούμε να κάνουμε από κοινού κατά τη διάρκεια του επερχομένου εξαμήνου και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Αναφερθήκατε στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα διαγνωστικά προϊόντα Μα ενδιαφέρει να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και ο δικό μου στόχο, όπω και ο δικό σα, θα ήταν να επιτευχθεί αυτό κατά τη διάρκεια του εξαμένου τη ε, Λουξεμβουργική προεδρία. Εάν δεν γίνει αυτό δυνατό, θα χρειαστούμε παρατάσει, αλλά θα ήταν καλό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το θέμα του λεγόμενου ελέγχου, σκρούτινη, είναι απαραίτητο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν να παρέμβουν αν υπάρχει, αν υπάρχει αμφιβολία σε σχέση με την κοινοποίηση για τα προϊόντα αυτά. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε το εξή. Είπε το Συμβούλιο ότι θα υπάρχει αυτή η διαδικασία δυνατότητα παρέμβασης αλλά μονάχα για μια μικρή ομάδα προϊόντων. Ενώ το Κοινοβούλιο στην δική του εντολή είχε την ε, λύση να περιλαμβάνεται ένας ευρύτερος χώρος προϊόντων και να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης μονάχα σε περίπτωση προβλημάτων. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι να γίνεται αυτή η διαδικασία όταν είναι απαραίτητη, αλλά να καλύπτει ένα ευρύτερο χώρο προϊόντων. Το να βρούμε μια συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά θα ήταν πολύ θετικό. Για τα διαγνωστικά προϊόντα, <clears throat> συζητήσαμε και προσωπικά, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην έννοια της συνένεσης μετά από πληροφόρηση του ασθενούς και επίσης για τους άλλους τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η κλωνοποίηση. Καταρχήν εδώ είναι σαφές ότι δεν είναι επαρκής η πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία η οποία να πλησιάζει περισσότερο και προς θέση του Κοινοβουλίου και ξέρω ότι το Λουξεμβούργο είναι πάντα ένα κοινοβουλιόστροφο έθνος και είναι φιλικό προς τις απόψεις του Κοινοβουλίου και θα μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες παραχωρήσεις. Τέλος για τα αντιβιωτικά <clears throat> θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ και εδώ όμω θέλω να επιστήσω την προσοχή σας για του, τα βακτήρια τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά και τα προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία, χρειαζόμαστε να δώσουμε κίνητα για την ανάπτυξη περαιτέρω αντιβιωτικών που δεν θα έχουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Ματίας Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Το θέμα της πρόσβασης στα ιατροφαρμακευτικά σκευάσματα μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί στο Κοινοβούλιο και την ιδίω τη δική μας πολιτική ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ιδίω με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τα σκευάσματα για την υπατήτηδα σε, το Κοινοβούλιο είχε κάνει μια ακρόαση για τα θέματα αυτά και είχαμε τονίσει επίσης και τη σημασία των διαμεθοριακών παροχών υγειονομικής περίθαλψης Έχετε λοιπόν πρόθεση να κάνετε κάτι το εξάμεινο της Προεδρίας σας για να βελτιώσετε το νομικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά, γιατί προς το παρόν όλα αυτά καλύπτονται από τις εθνικές ρυθμίσεις. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το νομικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις ανισομέρειες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. Και υπάρχει και το θέμα πολλές φορές της ε, έλλειψης προϊόντων σε ορισμένες χώρες για ορισμένα προϊόντα και εκεί θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει μια δυνατότητα να μπορεί κανείς να προσπορίζεται αυτά τα προϊόντα <clears throat> με διαμεθοριακό χαρακτήρα. Θα ήταν χρήσιμο, χρήσιμο λοιπόν να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια καλύτερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά. Η, αντί, η σε αντιβιωτικά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα επίσης του γλυφοσάτ είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Της γλυφοσάτης του παραστοκτόνου αυτού ο, στην δική μου περιοχή ε, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας ότι υπάρχουν σαφή δείγματα ότι παρουσιάζεται στον υδροφόρο ορίζοντα ίδρυ ίχνη γλυφοσάτης από το παραστοκτόνο Roundup. Επομένως και ο Πίτερ Λίζε αναφέρθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε νέες μορφές αντιβιωτικών και η κυρία Γκροστέπ επίσης αυτά που είπανε Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο να έχουμε μια νέα αντιμετώπιση για τα αντιβιωτικά. Δεν έχουμε λοιπόν άπειρο χρόνο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάσουμε όλες αυτές τις εκθέσεις για τα αντιβιωτικά. Χαίρομαι επίσης ότι η οδηγία για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται. Εμεί αναμείναμε πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω ότι και μέσα στο επόμενο εξάμεινο τουλάχιστον εν μέρη θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Κάτι ακόμα όμως πρέπει να σας πω για ένα τομέα που αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίων. Νομίζω ότι δεν κάνουμε επαρκή πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια σημαντική φάση στην ευρωπαϊκή πορεία και υπάρχει πολλές φορές πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν πιέσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα προηγουμένως, να σκεφτούμε περισσότερο για τις διαμεθοριακές παροχές ιατροφαρμακευτικής περίταξης. Έχουμε πάρα πολύ χώρο, και δρόμο να καλύψουμε, να ενισχυθεί περισσότερο αυτός ο διαμεθοριακός χαρακτήρας γιατί θα δώσει σε πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη να ξαναγίνουν <clears throat> υγιείς, να αντιμετωπίσουν ασθένειες με τη βοήθεια ιατροφαρμακευτικών ε, παροχών από γειτονικέ χώρε. Και έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα και ο ανταγωνισμό. Θα σα ήμουν ευγνώμων αν αναλάβετε το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε και στις στρατηγικέ με τις οποίες θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Εγώ απογοητεύτηκα όμως από την ε, Κομισιόν γιατί πολλές φορές έχει μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση θα ήταν καλό στον τομέα αυτό το Συμβούλιο να είναι ο σύμμαχός μας και να ασκήσει περισσότερο προς την Κομισιόν για να υπάρξει πρόοδο στα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι οι επόμενοι μήνες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Όπως προτείνεται είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνάπτουν και επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με τις δικές μας ε, ε, θέσεις του Κοινοβουλίου και περιμένω την απάντησή σας. Με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιέχα από τις μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα την ομιλία σας που ήταν διεξοδική. Αναφερθήκατε στις προτεραιότητες αλλά και σε κέρια ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά Μερικά πράγματα μου έλειψαν από την ε, ομιλία. Το Μάιο, τον, τον Μάιο στην Πολωνία είχαμε ε, περίπου 300 κρούσματα ε, σοβαρών ε, δηλητηριάσεων ε, εξαιτίας κάποιων ε, ψυχότροπων ουσιών. Και εδώ και καιρό σχολεί το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα αυτό. Ήδη τον Ιούλιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια σχετική έκθεση κα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην αγορά των νέων εντό εισαγωγικών ναρκωτικών, των νέων ψυχότερων πονοσιών είναι πολύ ανησυχητική και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Ε, τέσσερις προεδρίες διαδοχικές ε, ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, αλλά αποτέλεσμα ουδέν. Και ας δούμε τα στατιστικά του Ευρωβαρομέτρου. Ποιες είναι οι απειλές, ε, ποιος ο κίνδυνος των ανθρώπων που έχουν επαφή και χρησιμοποιούν αυτά τα θέματα. Στην Ιρλανδία, 42% 13% στην Αγγλία, 12% στην, ε, στην Γαλλία, στην Πολωνία 9%. Είχαμε όμως και ε, θανάτους από δηλητηριάσεις με τέτοιες ψυχότροπες ουσίες. Ερωτώ λοιπόν, η Προεδρία του Λουξεμβούργου ε, μήπως ξέχασε αυτό το θέμα. Ελπίζω όχι καλό θα ήταν και η Προεδρία του Λουξεμβούργου να συνεχίσει τις εργασίες ε, τεσσάρων προηγούμενων ε, ε, προεδριών που δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε συνένεση. Γιατί είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση με αυτά τα νέα ναρκωτικά, τις νέες ψυχότροπες ουσίες και θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση να ασχοληθείτε κατεπηγόντως με το θέμα αυτό. Πολλά δε μάλλον που έχουμε ελεύθερο εμπόριο και ε, αυτά τα νέα ναρκωτικά, οι νέες ψυχότροπες ουσίες, δεν είναι καν παράνομες, γιατί με, διαφορετικούς, με διαφορετικές ονομασίες και ε, διαφορετικές δραστικές ουσίες, νομότυπα διανέμονται στην αγορά, παρόλο που αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν ε, την φάση της διεκπαιρέωσης αυτών των εργασιών, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, θα πρέπει επιτέλους κάπου να καταλήξουν. Ελπίζω να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα στις προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, με τις οποίες κατά το λοιπού συμφωνώ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα, το λόγο έχει η κυρία Μέισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μούτς για την πλήρη της παρουσίαση. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, με βλέπετε, εδώ είμαι. Είναι πολλά αυτά τα οποία είπατε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα διεξέλθω όλα. Πολλοί συνάδελφοί μου ε, αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε μεταλαμπάδευση βελτί, ε, βελτίστων πρακτικών σε ό,τι αφορά την άνοια. <clears throat> Γιατί έχουμε μια κοινωνία η οποία γυράσκει και επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, η, όπως ελέγχθηκε από τον κύριο η διαμεθοριακή παροχή υγειονομικών ε, φροντίδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε και εσείς να δείτε πόσο έχει βελτιωθεί και αν έχει βελτιωθεί η κινητικότητα των ασθενών και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα από το Συμβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν για το γεγονός ότι σας ε, ενδιαφέρει και το θέμα αυτό. Ένα τρίτο ζήτημα είναι φυσικά οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Είπατε ότι υπάρχει εδώ μια πρόταση της Κομισιόν. Εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε πάντα επικριτικοί γιατί νομίζουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν αντιμετωπίζει και δεν επιλύει τα προβλήματα Βρισκόμαστε ακόμα στο, στο στάδιο της ε, συζήτησης, δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Τα, μου, τα ερωτήματα μου αφορούν την οδηγία για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. Εμείς περιμένουμε κατεπηγόντως να προχωρήσει το θέμα αυτό, όπως είπε και ο κύριος Λίζε. Και επίσης κάτι άλλο που αναφέρατε, ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα εξαρτάται από το Συμβούλιο το να προχωρήσει το θέμα των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Θα μπορέσουμε όμως να βρεθούμε σύντομα σε ένα τριγωνικό διάλογο για τα θέματα αυτά προς το καλό των ασθενών και ένας άλλος τομέας που με ενδιαφέρει είναι η <clears throat> καινοτομία υπέρ του ασθενούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε καινοτομία στα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και είναι επίση σημαντικό αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για όλους τους ασθενείς. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο. Ξέρετε ότι έχουμε μια οδηγία περί διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά έχει μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο και τελικά απεσύρθη από την Κομισιόν, δεν έχει προχωρήσει. Ενώ για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εργαστούμε περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ε, διαφάνεια. Υπάρχει μια διάσκεψη για τα θέματα αυτά τον Ιούλιο και το ερώτημά μου είναι κατά πόσο η πρόταση αυτή έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Υπάρχει δυνατότητα να την προωθήσετε στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθεί το θέμα αυτό. Μετά και από την απόσυρση της πρότασης από την Κομισιόν. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Όταν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε την χρήση των αντιβιωτικών, και πρέπει να δούμε πού θα μειωθούν ή μπορούν να αποφευθούν. Το ερώτημα είναι ποιε είναι οι εναλλακτικέ δυνατότητε που υπάρχουν. Αυτό μπορεί να είναι περιφερειακό θέμα για πάρα πολλού, αλλά υπάρχουν τα ζητήματα τη ομοιοπαθητική. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερη χρήση ομοιοπαθητικών και φυσικών ε, φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Απ' την ο κύριο Εκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, κυρία Μούτς που ήρθατε εδώ και μας τονίσατε ποια είναι τα κύρια θέματα που θα ενδιαφέρουν τη Λουξεμβουργική Προεδρία. Για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εσείς έχετε ε, αναφερθεί, συμφωνώ και είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει και ένα θέμα όμως το οποίο μου είναι ιδιαίτερα πρόσφυλες, είναι το θέμα των πολυανθεκτικών βακτηριδίων κάθε χρόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν 25.000 άτομα από τέτοιες πολυανθεκτικές μολύνσεις. Αποτελούν ένα, μια δαμόκλια σπάθα ένα, για την ε, ένα ξύφο του Δαμοκλή για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον πληθυσμό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολυανθεκτικές μολύνσεις ε, πολλές από αυτές προκύπτουν και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η, η γεωργία και η εκτινοτροφία όπου υπάρχει όλο και αυξανόμενη χρήση των αντιβιωτικών στη γεωργία και την εκτινοτροφία για λόγους προληπτικούς. Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι εναντίον της μαζικής αυτής χρήσης αντιβιωτικών και ιδίως της προληπτικής χρήσης στη Γεωργία. Θα υπάρξει λοιπόν κάποια κίνηση από την πλευρά του Συμβουλίου, θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για νομοθετική ρύθμιση και δεύτερον για το θέμα των ε, γενικά τροποποιημένων προϊόντων. Έχουμε όλο και περισσότερο εφαρμογή ε, ε, εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα. Για το κρέας του κουνελιού το 30% της κατανάλωσης στην Ευρώπη τώρα καλύπτεται από την ε, Κίνα και για την εκτροφή αυτών των ζώων υπάρχει μαζική χρησιμοποίηση αντιβιωτικών και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα που αναφέραμε προηγουμένως για τα αντιβιωτικά. Επίσης υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας το οποίο προξενείται για, από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκτροφή των ζώων στην ε, Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι κατά την Λουξεμβουργική Προεδρία και να κάνουμε κάτι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα. Να φύγουμε λοιπόν από μια εντατική ε, κτηνοτροφία και να προχωρήσουμε προς μια μορφή κτηνοτροφίας η οποία συμβάλλει στο να υπάρχουν πολύ λιγότερες ασθένειες στα ζώα αυτά με θετικές συνέπειες και για την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούρμες από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα, Λίδια. Χαίρομαι για το γεγονός ότι έχει κινητοποιηθεί η Λουξεμβουργική Προεδρία με ένα ευρύ και, θα, και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι η οδηγία για τις διαμεθοριακές παροχής περίθαλψης. Το Λουξεμβούργο βέβαια είναι η χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο αυτές τις δυνατότητες λόγω και της γεωγραφικής θέσης του. Έχουμε 108.000 άτομα από τον περίγυρο του Λουξεμβούργου που εργάζονται σε εμά και καλύπτονται από λουξεμβουργικά ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μπορεί να παίρνουν την περίθαλψη στο χώρο στις ε, στο χώρο κατοικίας τους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και κάποιον ε, απολογισμό για όλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία μεταξύ των ε, δικαιωμάτων των ε, ασθενών και των δυνατοτήτων περίθαλψης. Όλα αυτά φαίνεται ότι από την πλευρά της Κομισιόν οδηγούν σε μια ενκρυπτό φιλελευθεροποίηση τη παροχή περίθαλψης, αλλά η ασθένεια, η υγεία των ε, ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική για να είναι μοναχα αντικείμενο Επίση, Επίσης, ε, το πρόβλημα με τα εφητεύματα ασθήτους το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, οδήγησε σε αυτό το σκάνδαλο το οποίο αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα ήμουν ιδιαίτερα υπερήφανος αν η Προεδρία του Λουξεμβούργου μπορεί να δώσει μια ε, οριστική λύση στα προβλήματα αυτά. Ξέρουμε ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο το οποίο δεν υπήρξε η πολιτική θέληση για να αντιμετωπιστεί και βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει η πίεση των λόμπι να κουκουλώνονται όλα αυτά τα θέματα. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. και εμείς και πάλι γνωρίζουμε την νέα Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρχει η Προεδρία της Κομισιόν, θα υπάρξει μια δημοκρατική λήψη απόφασης για τα γενετικά τροποποιημένα και μετά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού με το Κοινοβούλιο από τη μια μεριά και την Προεδρία του Λουξεμβούργου από την άλλη πλευρά, ώστε να υποχρεώσουμε την Κομισιόν και τον κύριο Γιούγκερ τελικά να κάνει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Πρέπει να δημοκρατικοποιηθεί λοιπόν η διαδικασία λήψη απόφαση για του ιερατικά τροποποιημένου οργανισμού και πρέπει να τονίσω ότι εδώ η Κομισιόν είχε παρουσιάσει ε, 12 με 15 προτάσεις σε κάποιο έγγραφο, το οποίο έγγραφο δεν έχει δοθεί στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις να ασκήσουν πίεση στην Κομισιόν. Δεν μπορεί η Κομισιόν να προτείνει πράγματα μόνο σε εσωτερικά έγγραφα και να υπόσχεται να δώσει μια λύση και μετά να μην δίνει τα έγγραφα αυτά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδεχομένω. Τέταρτον, ένα από τα κυριότερα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σήμερα είναι ακριβώ η αντίσταση, η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να δούμε με την οδηγία για τα κτηνιατρικά φάρμακα ότι θα πρέπει ορισμένα αντιβιωτικά, με την οδηγία αυτή καταφέραμε ορισμένα αντιβιωτικά να αποσυρθούν από την κρίση στην κτηνοτροφία. Αυτό λοιπόν είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρώπη, επομένως και το Κοινοβούλιο και εσείς θα πρέπει να τα προωθήσετε. Γιατί χρειαζόμαστε να δώσουμε μια απάντηση στην αφεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο γίνεται αυτή η χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία οδηγεί σε άμεσους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Προεδρεύουσα και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία σας και θα είχα ένα σωρό ερωτήσει να κάνω κανονικά, αλλά θα επικεντρωθώ στο θέμα που εσείς αναφέρατε όσον αφορά την ε, εξατομικευμένη τα εξατομικευμένα φάρμακα, γιατί εγώ προέρχομαι από εκείνο το πεδίο και έχω παρακολουθήσει κάπως αυτή τη διαδικασία που καλεί να παράγεται όλο ένα και περισσότερο, να παράγονται όλο ένα και περισσότερο φάρμακα εξατομικευμένα. Η στόχη εντάξει, είναι ε, λογική και εγώ ίδιο συμμετείχα σε αυτή την επιστημονική ανάπτυξη ε, ε, ατομικών φαρμάκων. Όμως διαπιστώνω πως η μεθοδολογία αυτή ευνοεί τις φαρμακοβιομηχανίες και τις κατασκευάστρες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Γιατί εξατομικευμένη ιατρική σημαίνει ε, και εξατομικευμένες παροχές, παροχή, για το φαρμακευτικής περίθαλψης. Πολύ συχνά οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου είναι ελληματικές και αυτό πολλές φορές δεν αιτιολογείται από επιστημονική άποψη. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να οδηγήσουν σε τεράστιες δαπάνες που είναι, επιβαρύνουν τις δημόσιες ε, ε, τους δημόσιους οργανισμούς που και πάνε στις τσέπες των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών. Διερωτώ λοιπόν, τι μέτρα έχετε σκεφτεί να λάβετε ώστε να αποφύγετε τον πολλαπλασιασμό αυτού του τύπου των παροχών και άρα και την να αποφύγετε και την ε, υπερφόρτωση των υγειονομικών συστημάτων ενώ θα βελτιωθεί η παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Τώρα, σε περίπτωση πυρηνικής επίγουσης ανάγκης ή ατυχημάτων που μπορεί να προκύπτουν από κακή διαχείριση των ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων. Εσεί τι μέτρα θα λάβετε απέναντι στα κρατημέλη τα οποία δεν αναλαμβάνουν ε, τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ιδιαίτερα λόγω διαφθορά Και δίνω το παράδειγμα δυστυχώ τη Ιταλία που ακόμα δεν έχει εθνικό πρόγραμμα και παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει την φάση ε, εντοπισμού ενό συγκεκριμένου χώρου για την ταφή, για την ε, ε, των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Επελέγησαν οι συγκεκριμένοι χώροι με πολιτικές αποφάσεις, με καμία διαβούλευση με τον, και με το κοινό. Και αυτό είναι εις βάρος της υγείας, διότι η ανικανότητα, η διαφθορά και η πολιτική παρέμβαση έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των πολιτών. Τι θα κάνετε λοιπόν για να προλάβετε τέτοιου είδους υγειονομικές επίγουσες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Τελευταίος της, η κυρία Ντορνανό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Θα ήθελα ε, να ε, θίξω δύο σημεία τα οποία οποία δεν είναι στην πρότασή σας, αλλά που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά ε, και αυτό σημαίνει, ε, αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ιδιαίτερα στη γλυφοσάτη και το μαλάθιον που πρόκειται για ζενεκτόνα που έχουν ε, καταταγεί τον περασμένο Μάρτιο στην κατηγορία 2 2-1 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Δηλαδή, πιθανότατα καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Και ωστόσο όλοι κάνουν πως δεν ε, είδαν τίποτα. Η γλυφοσάτη, σας θυμίζω, είναι ένα από τα ζενεκτόνα που περισσότερο χρησιμοποιείται τόσο από τους γεωργούς όσο και από τους ιδιώτες. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα η Προεδρία του Λουξεμβούργου να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα υπέρ των ε, συμπολιτών μας. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ποιε είναι οι θέσεις σας ε, σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες άλλο σημείο που θέλω να θίξω είναι τα νανοηλικά. Οι επενδύσεις στον τομέα της νανοεπιστήμης είναι, με, είναι μεγάλες. Ωστόσο, η, ε, ο προπολογισμό που είναι αφιερωμένο στην έρευνα σε σχέση με την πιθανή επικινδυνότητα της νανοτεχνολογίας είναι ελάχιστος. Θα ήθελα να δω ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να... Ε, ε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των μεγάλων εταιριών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν επεκτατικούς ορισμούς όσον αφορά την νανοτεχνολογία ώστε να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερα έσοδα. Ωστόσο υπάρχει κόσμο που καταγγέλει τον κίνδυνο της νανοτεχνολογίας ε, όταν αυτή δεν, γίνεται σωστή, δεν είναι σωστό αντικείμενο διαχείρισης γιατί το μέγεθος των νανοηλικών μπορεί να διεισδύσει και μέσα από τα ε, ρούχα ε, στον ανθρώπινο οργανισμό δεν θα πρέπει να γνώμη αυτή την πραγματικότητα. ω μέλη αυτή τη επιτροπή, έχουμε το καθήκον να ενημερώνουμε και να προστατεύουμε. Ε, όσο προχωρούμε λοιπόν στην ε, κοινωνική τεχνική, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανοιχνευτούν συγκεκριμένα προϊόντα και φτάνουμε σε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Θα θα προβλέψετε λοιπόν σαφή και ξεκάθαρη ετικετοθεσία ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται για την παρουσία νανοηλικών. Επιθυμείτε να επενδύσετε στην επιστημονική έρευνα έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τους υγειονομικούς κινδύνους που αντιπροσωπεύουν αυτά οι νανοεπιστήμες. Σας ευχαριστώ. σε ευχαριστώ. Και τώρα, κυρία Υπουργέ, μπορείτε να έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ε, σας ευχαριστώ όλους σας για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που υποβάλατε. Πολλοί ευρωβουλευτές ε, μίλησαν ιδιαίτερως για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Και δικαίως, γιατί πρόκειται για ένα θέμα που εκρεμεί χρόνια ολόκληρα. Και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε τις εργασίες για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Λίζε, ο κύριος Γκρότε, αλλά και η κυρία Μάισνερ, μεταξύ άλλων, έθεσαν ερωτήσεις ε, ζητώντας ε, λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των ε, εργασιών μας. Σας είπα ότι ήδη έχουμε τους μερικούς γενικούς προσανατολισμούς. Είναι γενικοί οι προσανατολισμοί, γι' αυτό και χρήζουν κάποιες διευκρίνησεις, είτε σε επίπεδο αιτιολογικών σκέψεων, είτε σε επίπεδο τεχνικών ε, λεπτομεριών. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε αυτές τις γενικούς προσανατολισμούς μερικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας και κάποιες αιτιολογικές σκέψεις για να έχουμε ένα πλήρες πλέγμα προσανατολισμών που θα εγκρίνουν ε, οι Υπουργοί στο Συμβούλιο του Φθινοπόρου. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θέλουμε και επίσημη εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Ακούσαμε κάποια σχόλια για τις μέχρι τώρα συμβαστικές προτάσεις. Ο κύριος Λίζε μίλησε για τον έλεγχο, το σκρούτινι, Υπάρχει διάσταση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό, όντως. Ε, δεν υπάρχουν όμως ε, αντιφάσεις, ε, δεν υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Θεωρώ ότι η συμβαστική λύση ωφελεί τον ασθενή. Και αυτό και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το θέμα του ελέγχου, το σκρούτινι. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, οι συζητήσεις για τι αιτιολογικές σκέψεις ξεκίνησαν στις 6 Ιουλίου, ήδη έχει αρχίσει η προσπάθεια, στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Επί Λουξεμβουργικής Προεδρίας. Στις 22 Ιουλίου θα έχουμε τα συμπεράσματα και θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες τεχνικές ασυναρτησίες. Αυτές θα τι εξετάσουμε από τις 23 Ιουλίου και μετά. Βλέπετε ότι δεν θα ξεκινήσουν αμέσως οι διακοπές μας. Και μετά το καλοκαίρι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουμε την τεχνική εξέταση ώστε στις 15 Σεπτεμβρίου να υποβάλουμε το ενοποιημένο κείμενο στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις δύο νομοθετικές προτάσεις, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro. Και θα υποβάλουμε το συμβαστικό κείμενο για την υιοθέτηση των γενικών προσανατολισμών στις 5 Οκτωβρίου. Και φυσικά θα σας κρατούμε ενημερούς για την πορεία των εργασιών στο μέτρο που προχωράμε. Η πρώτη συνεδρίαση με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει σήμερα το απόγευμα μάλιστα. Ο στόχος μας ε, είναι πραγματικά η διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων πριν το Συμβούλιο Υπουργών της 8 η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η δεδηλωμένη μας πρόθεση και για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και αυτό το χρονοδιάγραμμα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε και γι' αυτό προτείνουμε τρεις τιμερείς διαλόγους μεταξύ των αρχών Οκτωβρίου και τελών Νοεμβρίου ή αρχών Δεκεμβρίου. Εκεί θα ασχοληθούμε κυρίως με πολιτικά θέματα, αλλά θα λάβουν χώρα και τεχνικές συνεδριάσεις παράλληλα με τη διαπραγματευτική διαδικασία. Το θέμα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι από τις ε, πρωταρχικές προτεραιότητες ε, της Λουξεμβουργικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά, πολλοί ευρωβουλευτές, για παράδειγμα ο κύριος Γκρότη, η κυρία Μάστερ, ο κύριος Εκ και ο κύριος Τούρμες, τόνισαν τη σημασία αυτού του θέματος, της μικροβιακής αντοχής. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Συμφωνούμε ως προς αυτό. Και η προσέγγιση μας προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ε, του τομέα της υγείας των ανθρώπων και της υγείας των ζώων. One Health. Μία υγεία έχουμε και γι' αυτό λαμβάνουμε υπόψη τη σημαντική συνεισφορά της Ιδανικής Προεδρίας του 2012 και θα συνεχίσουμε το έργο της. Το σχέδιο δράσης άλλωστε εκπνέει το 2016. Οπότε θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι εργασίες αυτές που είναι πολύ σημαντικές για μας να συνεχιστούν με ικανοποιητικό τρόπο και μετά το 2016. Και είμαστε υπέρ της συνεργασίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το θέμα της μικροβιοικής αντοχής και μετά το 2016. Είναι κέριο ζήτημα και για μας. Θέσατε συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, για τις ε, συγκεκριμένες ε, εργασίες και τα εγχειρήματα της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Θα έχουμε πολυσχηδή προσέγγιση. Για παράδειγμα, θα έχουμε μία διάσκεψη κτηνιάτρων. Μόλις έλαβα την πρόσκληση για την διεθνή διάσκεψη κτηνιάτρων με θέμα την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Η διάσκεψη αυτή θα λάβει χώρα στις 23 Οκτωβρίου. Αλλά θα έχουμε και άλλη σημαντική διάσκεψη της Διατλαντικής Ομάδας Εργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ίδιο θέμα, τη μικροβιακή αντοχή δηλαδή. Οργανώτρια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίτλος είναι να παραμείνουν αποτελεσματικά τα αντιβιωτικά. Και οι δύο εκδηλώσεις και οι δύο διασκέψεις θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο. Σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα ε, για την Προεδρία του Λουξεμβούργου και θα δώσουμε τη σκητάλη στη συνέχεια και στην Ολλανδική Προεδρία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες με τους συναδέλφους ε, για να συνεχιστούν ε, οι ενδιαφέρουσες αυτές ε, διαλέξεις και να δοθεί κάποια συνέχεια και μετά την βραδιά του Λουξεμβούργου. τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις και για ένα άλλο νομοθετικό θέμα, ζήτημα, τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Το μήνυμα ελήφθη. Κατάλαβα ότι περιμένετε από εμά και προσδοκάτε να προχωρήσουμε όσο γίνεται στο θέμα αυτό. Φυσικά δεν ξεχνούμε και θα παρακολουθήσουμε την ψηφοφορία που θα γίνει στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί η αναθεώρηση του κεκτημένου θα διευκολύνει την πρόσβαση στα κτηνιατρικά φάρμακα και θα μειώσει το γραφειοκρατικό άχθος σε επίπεδο καταχώρησης των φαρμάκων αυτών, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα, θα ενισχύσει την καινοτομία, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμβάλλει σε ενισχυμένη ασφάλεια του καταναλωτή. Εκεί θα επικεντρωθούν οι προσπάθειές μας ε, στις άδειε παρασκευής και διανομής που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ε, επίσης το θέμα της βάσης των δεδομένων και θα υποβάλουμε και πρόταση με θέμα τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλονται για τα κτηνιατρικά φάρμακα ή τις εισφορές. Αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα προς το τέλος της Προεδρίας μας. Δεν νομίζω να προλάβουμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση του κειμένου. Θα ήταν παραπλανητικό να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Πολλές ερωτήσεις ε, τέθηκαν και για την κλωνοποίηση. Και από τον κύριο Λίζε και από άλλους ευρωβουλευτές. Η Προεδρία μας προτίθεται να ξεκινήσει την εξέταση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τεχνικό επίπεδο. Γνωρίζω ότι έχετε αρχίσει την εξέταση των προτάσεων και επίσης γνωρίζω ότι γίνονται σφοδρές συζητήσει για τη νομική βάση. που αφορούν έμεσα και την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση των συζητήσεων. Άλλο σημαντικό θέμα αφορά την ετικετοθεσία των ε, προϊόντων ε, που προέρχονται από γόνους ε, κλόνων. Και ρωτήσατε αν θα προτείνουμε ειδικά μέτρα για την ε, θέση στην αγορά τροφίμων που προέρχονται από κλόνους ή γόνους κλόνων. Εμείς ε, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτές τις τεχνικές συζητήσεις και έχουμε την πρόθεση να αρχίσουμε την εξέταση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στα φάρμακα και το θέμα της ε, τιμής των φαρμάκων, της τιμολόγησης των φαρμάκων, το θέμα αυτό αφορά και τα καινοτόμα φάρμακα, αλλά και την ανταλλαγή απόψε, την ανταλλαγή ε, πληροφοριών Αυτό το θέμα απασχόλησε πολλούς ευρωβουλευτές της ομιλίες τους και μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου η Προεδρία μας θα συνεργαστεί με το επόμενο τρίο Προεδριών, δηλαδή τις κάτω χώρες, τη Σλοβακία. Που αποτελούν την επόμενη επερχόμενη τρόικα Προεδριών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μια συζήτηση στην ομάδα Δημόσιας Υγείας η οποία συνεδρίασε χθε εξάλλου και προσπάθησε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα αυτά. Επομένως και ως εκ τούτου έχουμε πράγματι ξεκινήσει τις εργασίες μας και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μεν ανεπαρκείς πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο του Συμβουλίου αλλά πολλά κράτη-μέλη έχουν υποστηρίξει το κείμενο παρά το γεγονός ότι άλλα κράτη-μέλη αντιστάθηκαν στο κείμενο αυτό. Πιστεύω λοιπόν κατά την άποψή μου ότι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά την απόφαση, τις αποφάσεις για την τιμολόγηση των φαρμάκων από τα κράτη-μέλη και τις αποδόσεις τους ασθενείς και επίσης τον τρόπο με τον οποίο η φαρμακευτική βιομηχανία καθορίζει τις τιμές ώστε συνολικά να μπορέσουμε να μειώσουμε τις τιμές. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η τιμολόγηση σε ό,τι αφορά ε, τις επιστροφές προς τους ασθενείς του κόστους των φαρμάκων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κάθε αλλά κατά την άποψή μου ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά είναι η εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών για τα διάφορα μοντέλα τιμολόγησης και απόδοσης εξόδων στα κάτι μελη και η συμμετοχή εθελοντικά βέβαια της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αλλιώς δεν θα έχουμε καμία πρόοδο. Χαίρομαι για αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά την πολιτική για το αλκοόλ. Εμείς θελήσαμε αυτό να είναι ένα βήμα για μια συζήτηση και έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση της Κομισιόν για την ε, ε, ε, σήμανση σε ό,τι αφορά την θρεπτική αξία των αλκοολούχων ποτών. Είναι λοιπόν πολλές πτυχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η κοινωνική πτυχή, η οικονομική πτυχή σε ό,τι αφορά την κατάχρηση αλκοόλ, αλλά φυσικά και η πτυχή της δημόσιας υγείας και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να έχουμε μια συνεργασία διαμεθοριακή για τα θέματα αυτά και κυρίως ότι αφορά και την διαφήμιση και τις πωλήσει στο διαδίκτυο και τις επιρροές που μπορεί να έχουν αυτές οι βλαβερές συνήθειες για τους νέους. Για τον κύριο Πέισα είχε τονίσει επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα αλκοολούχα ποτά, αλλά αναφέρθηκε και στις νέες ψυχοτροπικές ουσίες σε σχέση με την πολιτική αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Τώρα υπάρχει η οριζόντια ομάδα ναρκωτικών στην, ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης. Ξέρετε όμως ότι αυτό άφτεται θεμάτων δημόσιας υγείας και φυσικά το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί σε συνάρτηση με όλα τα θέματα της υγιεινής ζωής, του υγιεινού τρόπου ζωής που υποστηρίζουμε αλλά το θέμα αυτό, αυτό κάθε αυτό εκφεύγει της αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής και φυσικά και των δικών μου καθηκόντων ως Υπουργού Υγείας. Αλλά είμαι σε επαφή με την ομόλογο μου Υπουργό Δικαιοσύνη ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συναρμογή των πρωτοβουλειών στον τομέα αυτό για την αντιμετώπιση των θεμάτων λοιπόν δημόσιας υγείας. χαίρομαι ιδιαίτερα και για τις θετικές σας ε, αντιδράσεις σε σχέση με το θέμα της ε, άνοιας. Αυτά που είπε η κυρία Μάισλερ βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια εναρμόνιση των διαφορετικών πολιτικών σε σχέση με την άνοια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διαμεθοριακές συνεργασία στον τομέα αυτό, αλλά η άνοια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν και από την πλευρά των κυβερνήσεων πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις και οι ειδικέ ανάγκες των ανθρώπων αυτών που πλήττονται από αυτή την ασθένεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο περιγυρός τους και οι οικογένειές τους και την ανάγκη να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό της πολιτικής μας και της δράσης μας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμερίζομαι απόλυτα όλα αυτά τα οποία αναφέρατε για το θέμα αυτό. Επίσης, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. «25 χρόνια είμαι κοινοβουλευτικός στη χώρα μου, οπότε ξέρω πόσο ενδιαφέρονται τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μονάχα τους Υπουργούς Υγείας, αφορά όμω και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, τους Υπουργούς Γεωργίας και έχετε ορθά υπογραμμίσει τη σημασία που έχει η συζήτηση του θέματος αυτού σε σχέση με τις διάφορες πολιτικές για τον τομέα της γεωργίας, της πρόληψης ασθενειών, του περιβάλλοντος. Επίσης και αυτό αναφέρθηκε από τον κύριο Εκ. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει βέβαια την πρόταση αυτή και προβλέπεται να υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αυτά. Εγώ... Και διαπιστώνω ότι τα όσα λέτε εσείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι παρόμοια με τις ε, επικρίσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και ε, ε, τις επικρίσεις και τις απόψεις διαφόρων υπουργών και ότι έχετε την Μπορώ να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε διακόπτη ο Πρόεδρος γιατί χρειαζόμαστε χρόνο για να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Άλλωστε θα κάνουμε συστάσεις λοιπόν στο θέμα και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ. Θα έχω πολλές ερωτήσεις να σας θέσω κυρία Υπουργέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν, εξατομικευμένη ιατρική. Είναι το μέλλον αυτό. Και πιστεύω πως αυτού του είδους ιατρική θα βρει τον τρόπο να θεραπεύσει ε, ασθενείς που ακόμα δεν να μπορούν να θεραπευθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί και η υγεία, η ηλεκτρονική υγεία και ξέρετε ότι εκεί το μπλοκάρουν τα κράτη-μέλη και αυτό το ζούμε μέσω της εφαρμογής ε, της, διασυ... της οδηγίας περί διασυνοριακών ε, ιατρικών αγωγών, ιατροφαρμακευτική περιθαψη Εν πάση περιπτώσει, η εφαρμογή τη δεν είναι ικανοποιητική. Είπατε ότι θα κάνατε με έναν απολογισμό, αλλά στην πράξη πρέπει πραγματικά να γίνει κάποια δράση προ τα κάτι μέλη, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική ε, ε, και επιχειρησιακή. Η θέληση που έχετε να δούμε το μέτρο της εναρμόνισης και της κεντρικής ε, ανάλυσης κόστους ωφέλους των νέων φαρμάκων που γίνονται αυτή τη στιγμή μεμονωμένα σε κάθε κράτος μέλος. Ξέρω πως η Κομισιόν είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και αυτό σημαίνει πραγματική βούληση από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να έχω τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Η Άνια, είμαι πρόεδρος εδώ και 8 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ασθένειας της, του Αλτσχάιμερ. Ε, είμαι ευτυχής που είναι προ, ε, προτεραιότητά σας η Άνια. Θα ήθελα ε, ε, να σας πω ότι ωστόσο για την Αλσχάιμερ δεν γίνονται τόσα πράγματα ε, και είναι άνηση η κατάσταση στα κρατημέλη. Ποια είναι η άποψή σας και τι θα κάνετε γι' αυτό. Τώρα, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Συμφωνούμε όλοι στο Κοινοβούλιο για να καταπολεμήσουμε την αντίσταση στα, μικροβια... στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό σημαίνει απόλυτη αγόρευση της προληπτικής χρήσης των αντιβιωτικών και πρέπει επίσης να ρυθμιστεί η πώληση στο ίντερνετ. Δηλαδή ε, να απογορευτεί από τη μια πλευρά η πώληση των αντιβιωτικών και ίσως και όλων των φαρμάκων που δίνονται μόνο με ε, συνταγογράφηση. Ήθελα να σας μιλήσω και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η Κομισιόν φρενάρει όσο μπορεί σε αυτό το θέμα. Θα ήταν καλό το Συμβούλιο να δράσει ώστε να προχωρήσει ο προβληματισμός στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ζιλ Παγνιό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα της κύρωσης ε, της σύμβασης του ΠΟΕ για το παράνομο εμπόριο ε, καπνού. Ε, από τότε έχω δημιουργήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια άτυπη ομάδα εργασίας κατά της παράνομης παρέμβασης της βιομηχανίας του καπνού. Συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες, ε, όλες οι εθνικότητες καθώς και εκπρόσωποι των συνδέσμων κατά του καπνίσματος. Η φιλοσοφία της ομάδας μας είναι απλή. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική κατά του καπνού, του καπνίσματος που στόχο έχει τους κατασκευαστές ε, προϊόντων καπνού και θέλουμε να ενθαρρύνουμε ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη και την Ένωση να κυρώσει αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας του ΠΟΕ που στόχο έχει να καταργήσει το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού. Μόνο 58 κράτη στον κόσμο για την ώρα έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο. Μεταξύ αυτών είναι η Ένωση στις 20 Δεκεμβρίου του 2013. Μόνο 8 την έχουν κυρώσει όμως από τα 58 που την έχουν υπογράψει. Δεν έχει ακόμα υπογράψει ούτε το Λουξεμβούργο μεταξύ αυτών. Οπότε ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών και δεδομένες προεδρία το Λουξεμβούργο θα υπογράψει αυτό το πρωτόκολλο. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε στη διάρκεια αυτών των έξι μηνών ώστε να επιτρέψετε όχι μόνο την υπογραφή από πλευράς της Ένωσης αυτού του πρωτοκόλλου συμφωνίας, αλλά επίσης να επιτρέψετε κατά αυτόν τον τρόπο να ε, διευκολυνθούν τα κράτη-μέλη που ακόμα δεν έχουν κυρώσει ε, υπογράψει ούτε κυρώσει αυτό το πρωτόκολλο. Δεύτερο σημείο είναι οι ενδείξεις προέλευσης για το κρέας για τα έτοιμα πιάτα. Ε, ξέρετε ότι έχουμε κάνει νέο ψήφισμα που ζητά την ε, υποχρέωση ετικετοθεσίας για το κρέας που χρησιμοποιείται στα μεταποιημένα προϊόντα. Ε, σε πρόσφατη δε συνομιλία με τον κύριο Ντρουκάιδη τον Ευρωπαϊκό Πίτροπο, δυστυχώ μου είπε ότι καμιά ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είχε προβλεφθεί μέχρι στιγμή. Οπότε και εδώ θα ήθελα, να, αν μπορείτε, να μας διευκολύνετε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. τελευταία παρατήρηση. Είπατε πριν από λίγο πως επιθυμούσατε την οργάνωση μιας διάσκεψης σε σχέση με την έμπολα. Εγώ στην προηγούμενη θητεία ήμουν εισηγητής για το ψήφισμα και την απόφαση για την ε, καταπολέμηση της, των ε, απειλών των διασυνοριακών για την υγεία και γι' αυτό και θα ήθελα να συμμετέχουμε σε αυτή τη διάσκεψη δεδομένου ότι η προστεθέμενη αξία αυτή τη απόφαση ήταν εξαιρετικά υψηλή στην καταπολέμηση του έμπολα, του ιού έμπολα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και την Υπουργό για τις ε, διευκρινήσεις που μας έδωσε. Εγώ θα ρωτούσα για το κρέας αποκλεινοποιημένα ζώα, αλλά ήδη απάντησε. Ε, το Κοινοβούλιο εμένει στην αρχική του θέση και αυτό φαίνεται και από τις τροπολογίες. Το Συμβούλιο θα αλλάξει γνώμη ή θα εμείνει και εκείνο στη θέση του. Γιατί ε, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, όπως συνέβη και στην προηγούμενη περίπτωση. Ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ηλεκτρονική υγεία, όπως ρώτησε η κυρία Γκροστέτ. Στην έκθεση πρωτοβουλίας μας ήδη θίξαμε τα βασικά προβλήματα, που είναι τα λειτουργικά συστήματα, τα επιχειρησιακά συστήματα και τα δικαιικά συστήματα για την αποδοχή ή τη συγκατάθεση των ασθενών. Εμείς έχουμε αποκεντρωμένες υπηρεσίες υγείας και σχετικές αρμοδιότητες και πιστεύω ότι χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, τι γίνεται με την κινητικότητα ε, υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τα κινητά και κανένα έλεγχος. Σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή περίθαλψη, πολύ καλή πρόταση, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το εύρος των υπηρεσιών, αλλά και η κοστολόγησή τους και αυτό σε συνάρτηση με την ηλεκτρονική υγεία. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, θα σταματήσω εδώ, αλλά η υγεία πραγματικά είναι ευρύτατο ζήτημα και πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κυρία Λίλενα Μπόρζαν. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που σας βλέπουμε στη συνεδρίασή μας ε, και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Προεδρίας σας που μας παρουσιάσατε. Επίσης, έμεινα ικανοποιημένη ε, και με αυτά που είπατε για τη στρατηγική για το αλκοόλ της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, γιατί μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει γίνει. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro, είμαι σκιώδη συγγήτρια για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σημειώσουμε πρόοδο στις σχετικές συζητήσεις. Το σχόλιο μου είναι ότι η η υγεία είναι εθνική ε, και ε, αρμοδιότητα και κάθε ε, κράτος κάνει τις επιλογές του ανάλογα με τις δυνατότητές του. Στην πράξη όμως φάνηκε ότι η υγεία έχει και διασυνοριακό χαρακτήρα. Ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό και κάποιες λύσεις θα πρέπει να τις βρούμε σε κοινοτικό επίπεδο. Και η οδηγία για τον καπνό ήταν ένα καλό παράδειγμα το πώς μπορούμε να βρούμε και οφείλουμε να βρούμε κάποιες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη σας, γιατί πρόσφατα ο Επίτροπος Ανδριοκάητες είπε ότι αν αλλάξει η συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνει μεταφορά των αρμοδιοτήτων της υγείας για πολλά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων για την υγεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εγώ ήθελα να θέσω εκ νέου μια ερώτηση που σας υπευλήσει ήδη, αλλά για την οποία ακόμα δεν λάβαμε απάντηση και αφορά τη γλυφοσάτη, την ε, ενεργή ουσία που χρησιμοποιείται περισσότερο στα ζυζανιοκτώνα. Από τη στιγμή που ε, δηλώθηκε ότι αυτή η ενεργή ουσία είναι μάλλον ε, ε, καρκινογόνος και τώρα περιμένουμε να, ε, να εκδοθεί αυτή η πλήρης έκθεση για αυτό το υπόθεση μέσα στο μήνα, πέρα που έχουμε και επιστημονικές ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι αυτή η δραστική ουσία είναι βλαβερή για την υγεία και για το περιβάλλον και αναφέρομαι στις αποκαλύψεις συγγνώμη, στην ύπαρξη αυτού, του, αυτής στα ούρα και στο ο, μητρικό γάλα. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση λοιπόν, δύσκολη και πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Ορισμένα κατημέρια έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση αυτής της δραστικής ουσίας, άλλοι ετοιμάζονται να το κάνουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν και εσείς ως Προεδρία σκοπεύετε κάτι να κάνετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταίο θέμα. Θέλω να ρωτήσω επίσης ότι αυτή την εβδομάδα ε, πήραμε στην Επιτροπή Αναφορών ε, τούντες ε, από, που είναι θύματα αυτού του φαρμάκου που από την δεκαετία του 50 έχει κάνει πολλά θύματα για τη θαλιδομίδη και έχει καταστρέψει τη ζωή τους. Πολλοί από, αυτά, από αυτούς δεν έχουν λάβει ποτέ αποσημειώσεις, ούτε καν έχει αναγνωριστεί ότι είναι ανάπηροι ε, υποφέρουν από αυτό και ζουν έτσι είναι εθνικό θέμα ε, της Ιταλίας αλλά με όλη, με, την, με όλη την ε, απαλή δύναμη και την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θέλω να ρωτήσω αν το Συμβούλιο σκοπεύει να κάνει κάτι για αυτή την φαρμακευτική τραγωδία. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σε σχέση με την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη ιατρική, ιατρική φυσικά δεν μπορώ να προκαταλάβω τα συμπεράσματα τα οποία θα ε, προέλθουν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα όμως όπως και για σας είναι ότι οι καινοτόμες θεραπείες να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κλινική πρακτική και μα, μου είπατε να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες για τις προκλήσεις αυτές. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των καινοτόμων φαρμάκων και της εξατομικευμένης ε, ιατρικής αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι όπως είπατε είναι πολλαπλού χαρακτήρα και γι' αυτό οι προσπαθειές μας εγγράφονται στα πλαίσια των συμπερασμάτων της ε, Ιταλικής Προεδρίας και η επικείμενη Ολλανδική Προεδρία και αυτή θα δώσει έμφαση στην πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της και έχουμε λοιπόν επομένως την εγγύηση να έχουμε μια μακροχρόνια ατζέντα. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Σημαίνει με την αποψή σας ότι είναι κατεπίγον να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κριτήρια σαφή που να αναφέρονται στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μια ανάλυση αντικτύπου θα πρέπει να μπορέσει να περατωθεί μέχρι τα μέσα του 2016 σε ό,τι αφορά τη γλυφοσάτη. Εμείς περιμένουμε την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και την ε, αξιολόγηση της ΕΦΣΑ σε σχέση με το προϊόν αυτό για τα νανοηλικά και τα νέα τρόφιμα. Χαιρόμαστε για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε τον Ιούνιο ήταν πραγματικά ένα σαφές και στεναρό μήνυμα και με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι εξυγχρονισμένο <clears throat> και που θα προσδώσει μεγάλο επίπεδο ασφάλειας για τα ζώα. Σας προσκαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη την δυναμική αυτή που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμανση, αιτή και τοθεσία των ε, τροφίμων. Είχατε αναφερθεί και στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων τον Δεκέμβριο του 2013 και τον ίού και το Μάιο του 2015 η Κομισιόν προετοίμασε εκθέσεις σε σχέση με το εφικτό μιας υποχρεωτικής σήμανσης για την χώρα προέλευσης και του τόπου προέλευσης για τα διάφορα τροφιμικά προϊόντα, ιδιαίτερα το κρέας, όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό το γάλα, το είδος του κρέατος, πέραν του βοηού κρέατος, του χειρίου κρέατος, του αιγίου και προβίου κρέατος και του πουλερίου κρέατος και επίσης των μεταποιημένων προϊόντων που έχουν ένα μονάχα συστατικό ή ένα συστατικό που εκπροσωπεί πάνω από 50% του τροφιμικού προϊόντος και στο φως των πορισμάτων των μελετών που έγιναν <clears throat> όταν υπάρχει υποχρεωτική σήμανση προέλευσης αυτό θα είναι ιδιαίτερα πολυδάπανο η Κομισιόν έχει ε, θέσει και μια νομοθετική πρόταση αλλά όπως ξέρετε τον Μάρτιο το Συμβούλιο έκανε μια ανταλλαγή απόψεων <clears throat> σε σχέση με την έκθεση για την ένδειξη προέλευσης και των συστατικών και τα κράτη-μέλη είχαν απόψει τελείως αποκλίνουσε σε σχέση με το εφικτό και το σκόπιμο της υποχρεωτικής ετικετοθεσίας. Η Κομισιόν λοιπόν παρουσίασε τα συμπεράσματά της στο Συμβούλιο σε σχέση με τα άλλα προϊόντα και οι πρώτες ε, αντιδράσεις των κατών μελών ήταν ιδιαίτερα ποικίλε τόνισαν τη σημασία να υπάρχει σωστή πληροφόρηση αλλά να αποτραπεί η δημιουργία πρόσθετου κόστους. Είναι δυνατή η εθελοντική αναφορά ε, της προέλευσης όσο δεν είναι παραπλανητική και όσο προέρχεται πραγματικά από τον παραγωγό των προϊόντων αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Υπουργό Μους για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Very interesting. Yes. <laughs> Dear colleagues, we have uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μέση διάταξη που είναι η έκθεση πρωτοβουλίας για μια νέα συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι με εισηγητή τον Γιλ Παρνιό. 230 τροπολογίες έχουμε. Πρωτού ξεκινήσω και δώσω το λόγο στον κύριο Παρνιό θέλω να ζητήσω όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν ησύχως και ηρέμως. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Γιλ Παρνιό για να παρουσιάσει την θέση του για τις τροπολογίες. Παρακαλώ, ησυχία. Συνεχίζουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε... 6 Ιουνίου την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή και εκεί σας παρουσίασα τα βασικά στοιχεία της έκθεση μου για την COP21 και κατέγραψα τις πρώτες αντιδράσεις. Στο μεταξύ Πολλοί καταθέσατε τροπολογίε επί της εκθέσεω. 230 τροπολογίε κατατέθηκαν στι 17 Ιουνίου 72 οι σοσιαλιστές, 48 το ΕΛΚ, 26 οι φιλελεύθεροι, 23 η ΣΥΑΡ, 18 οι πράσινοι, 17 μέχρι στιγμή η εγγεγραμμένη και 14 η 12 η ΓΚΟΕ. Να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεσή μου περιορίζεται από τους 8.000 8.000 ψηφία είναι δυστυχώ ε, πολύ σύντομη για ένα τόσο κέριο ζήτημα όπω οι κλιματικέ αλλαγέ. Γι' αυτό κατέθεσα και εγώ 34 τροπολογίε, ε, είτε μόνο είτε από κοινό με τους σοσιαλιστές ε, δημοκράτες, ώστε να αναπτύξω πιο διεξοδικά κάποιε πτυχέ τη έκθεσης. Οι τροπολογίε αυτές αφορούν την καταπολέμηση της αποψήλωσης, η διαδικασία κύρωσης των τροπολογιών της Ντόχα, το θεματολόγιο παράλληλων λύσεων μετά τη Συμφωνία του Παρισ, των Παρισίων, ώστε ε, οι κυβερνήσεις, οι πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να αποδείξουν ότι δεσμεύονται όντως ε, υπέρ της μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλή χρυσή άθρακα. Χθε είχαμε ανταλλαγή απόψεων και για τη μεταρρύθμιση του συστήματο εμπορία εκπομπών και των ποσοστώσεων του άνθρακα και έχουμε και κάποιε ιδιωτικέ πρωτοβουλίε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Με την σημερινή συζήτηση θα μπορέσει ο καθένας να παρουσιάσει τις τροπολογίε του και ευχαριστώ εκ των προτέρων τους και οδησηγητές και γενικώ τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Πάντως η πλειοψηφία των τροπολογιών ε, εμπλουτίζει την έκθεση και τη βελτιώνει. Και διαπιστώνω μια σύγκληση απόψε. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες για το σύνολο των θεμάτων. στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ και σε επιμέρους ζητήματα. Προτιμώ τώρα να ακούσουμε τους και ηγητές και τους ε, λοιπούς συναδέλφους για να μας παρουσιάσουν τις τροπολογίες τους. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Φλόρεντς από το ΕΛΚ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Να πω εξ αρχής ότι η συζήτηση για τη διάσκεψη του Παρισιού στο τέλος του έτους. Έγινε σε επίπεδο αντικειμενικό και συναδελφικό, κάτι το οποίο δεν γινόταν πολύ συχνά στο παρελθόν. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά που λέει ο συγητής, αλλά μου αρέσει η προσέγγιση του. Μπορώ να υποστηρίξω πολλά από αυτά τα οποία λέει. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κοινού δρόμους στο μέλλον και κυρίες και κύριοι. Είναι κάτι που πρέπει να το επαναλάβω. Είμαστε ισχυροί μόνο όταν έχουμε μια κοινή στάση και όταν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και με την Κομισιόν. Υπάρχουν κάποιες διαφορές σε αριθμητικά στοιχεία, το ξέρω, αλλά όταν εμείς εκπροσωπούμε τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών με ένα θετικό τρόπο μπορεί να έχει βάρος η άποψή μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε εσωτερικές διαμάχες για θέματα λεπτομεριακά όπως είναι το, οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση ή για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα διεθνές <clears throat> ε, πακέτο λύσεων και πρέπει εμείς ως Ευρώπη να είμαστε ενωμένοι. Είδαμε ότι πριν από μερικά χρόνια δεν έλαβε κανείς υπόψη τη θέση της Ευρώπης γιατί δεν θεωρούσαν ότι ήταν εφικτή και πρακτική. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και χαίρομαι για το γεγονός ότι και ο εισηγητής μας έχει θέσει προτάσεις οι οποίες πιστεύω ότι μπορούν να συνενώσουν όλοι μα, όλους μας ώστε μαζί με την Κομισιόν και τα κάτι μέλη να τις υποστηρίξουμε. <clears throat> Θέλω να πω κάτι εν συντομία για την χρηματοδότηση. Έχει εντωμεταξύ αποφασιστεί ότι όχι μονάχα να πληρώνουν οι βιομηχανικές χώρες, αλλά και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει και αυτές να συμβάλλουν. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Ούτε η Σαδική Αραβία ούτε και η Κίνα μπορούν να θεωρούνται πια ότι είναι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πιο δίκαια κατανομή βαρών και να υποστηρίξουμε το να παίξουν και αυτές οι, οι χώρες αυτό το ρόλο. Για δεν ξέρω για εσάς τη Γαλλία κύριε Παρνιό, αλλά για τη Γερμανία είναι δύσκολο να πείσουμε τον πληθυσμό να αναλάβει χρηματικά, χρηματοοικονομικά βάρη για την στήριξη συμφωνιών όπως αυτής του Παρισιού. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη κατανομή του οικονομικού βάρους και δεν μπορούμε να, να πιστεύουμε ότι μπορούν τα κράτη μας να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Όταν γινόταν η επανάνωση της Γερμανίας είχαμε πει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Γερμανίας θα μπορούσε να τα λύσει όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, χωρίς ιδιωτικό κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Αλλά φυσικά αυτό μπορεί να γίνει η συμμετοχή του ιδιωτικού και κεφαλαίου μόνο με σαφείς και δίκαιους κανόνες, όχι με αρπακτικούς κανόνες. Αλλά χωρίς ιδιωτικό κεφάλαιο δεν μπορεί να γίνει τίποτα τέτοιο, να προχωρήσει τίποτα. Και βλέπω, στρέφομαι και προς τους φιλελεύθερους, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της αγοράς αλλά <clears throat> πρέπει να έχουμε και ένα νέο οδικό χάρτη, ο οποίο να περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Προτείνει <clears throat> ο εισηγητή τον φόρο συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Δεν είσαστε μόνο σα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενιαίου ευρωπαϊκού κανόνε θα πρέπει να καταλάβουμε παρά το γεγονός ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε σε αφηρημένο επίπεδο αυτόν τον φόρο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος και δεν υπάρχει ε, συνένεση γι' αυτό, θα καταρρεύσει αυτή η προσπάθεια. Μάλλον είναι καταδικασμένη για αποτυχία αυτή η πρόταση, το βλέπω και από τη χώρα μου η οποία δεν νομίζω ότι έχει καμία θέληση προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να βρούμε πιο εφάνταστες λύσεις. Πιστεύω βέβαια ότι είναι σωστό να συζητήσουμε και εγώ χαιρετίζω την ε, αισιόδοξη στάση του εισηγητή και τέλος υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν δει το θέμα αυτό με θετικό τρόπο και το λέω αυτό σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι να βρούμε μια λύση στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρώτο. Ο κύριος Χερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παρνιό και τον κύριο Φλόρεντς για τις ε, πολύ ε, στεναρές τους ε, συμβολές σε αυτή τη συζήτηση μέχρι τώρα. Πιστεύω πως η σχέση με την κόπα είναι πολύ ισχυρή έκκληση προς την ομάδα σας, όντως. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι εγώ βλέπω κάποιες θετικές εξελίξεις Η Άντζελα Μέρκελ έδειξε πολλές ηγετικές, ε, έκανε μάλλον ε, ε, ολόκληρη παράσταση ηγετικής ικανότητας στο G7 και είναι πολύ θετικό αυτό στην πορεία για το Παρίσι, αλλά επίση βλέπω ότι υπευλήθη από την Κίνα, η οποία επιτέλους φαίνεται να αναλαμβάνει τις ευθύνες της την υπόθεση του κλίματος, όχι μόνο αντιπροσωπεύοντας την ομάδα των 77, αλλά και προσπαθώντας να κινηθεί πιο γρήγορα από, από άλλοτε. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε στο σωστό τους επίπεδο της δεσμεύσης της. Κάποια στοιχεία που θέλω να τονίσω στο δικό μας ψήφισμα. Καταρχήν, η σημασία της προστασίας των δασών. Ε, ανεφέρθη από άλλους σε παλιότερες συζητήσεις, ανεφέρθη ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης των σκιωδών που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Είδαμε ε, τροπολογίες που προήλθαν από διάφορες πλευρές του σώματος Οπότε θα ήταν ε, σπουδαίο αν μπορούσαμε να βρούμε μια έντονη διατύπωση από αυτού. Εγώ ίδιος έχω καταθέσει τροπολογία μαζί με τον συνάδελφο Φέντερλι. Ελπίζω λοιπόν πως θα βρούμε μια ισχυρή και φιλόδοξη συμβιβαστική εδώ. Δεύτερο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι η ικανότητα να χρηματοδοτηθεί πολιτική παγκόσμια εμβέλεια για τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω ότι αν έχουμε περισσότερο χρήματα από τους δημόσιους προπολογισμού, είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε αν και είναι απαραίτητο να γίνει από την πλευρά των πλουσιωτέρων αυτού του κόσμου αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα των αγορών άνθρακα όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που συλλέγονται εκεί ώστε να χρηματοδοτήσουμε προσαρμογές ε, στον άνθρακα και σε άλλα μέρη του κόσμου και είδα διάφορες τροπολογίες ε, από το ΕΛΚ, από τους σοσιαλιστές και άλλους και εκεί θα ήταν καλό να βρούμε συμβιβαστική. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι χρησιμοποιούμε δημόσιο χρήμα για να ε, δώσουμε πιστώσεις για εξαγωγές ε, τεχνολογίας ε, χρησιμοποιούμε δημόσια χρήματα για να εξασφαλίσουμε αυτές τις επενδύσεις, ας πούμε τεχνολογία ε, στην Κίνα, στην Ινδία και αλλού. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Οι πράσινοι ήδη έχουν πει ότι θα το στηρίξουν αυτό. Τι θα πρέπει να κάνουμε από σήμερα μέχρι το 2020 εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι στόχοι μέχρι το 2020, αλλά αυτό που είναι ε, σκόπιμο είναι να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ενημερώσει τον υπόλοιπο κόσμο για τα καταπληκτικά υπερεπιτεύγματα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Ότι δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τους ίδιους μας τους στόχους για το 2020 Είναι πολύ ισχυρό μήνυμα. Αυτά, Πρόεδρε. Και προβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στον εισηγητή κύριο Παρνιό και του Σκιώδη. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάβορ. Γιάβορ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης του που μας διευκολύνει γιατί επικεντρώνεται στα ουσιώδη σημεία που μια τέτοια έκθεση πρέπει να περιέχει. Πριν επισέλθω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σταθώ λίγο στον πιθανό στόχο μιας τέτοιας έκθεσης ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, και οι συμφωνίες θα γίνουν στο Παρίσι στα τέλη του έτους. Αυτό που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να στείλει ένα χειρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλους τους διαπραγματευτές, σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη για το ποια είναι η δική μας σκοπιά για τις κλιματικές αλλαγές και ποιε είναι οι προσδοκίες μας από τη διάσκεψη κορυφής των Παρισίων για το κλίμα. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι σημαντικό να διατρανώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ε, πρόδρομος ε, σε θέματα κλιματικών αλλαγών και κλίματος ε, και είχε ηγετικό ρόλο μεταξύ των θεσμικών οργάνων που θέλει να τον διατηρήσει. Ακόμη και ε, ως προς τους στόχους ε, Του αριθμού και τα ποσοστά που περιλαμβάνει η έκθεση και αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ηχηρού μηνύματος προς τους εταίρους ε, εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση, επαναλαμβάνω, έχει πολύ καλές προτάσεις και μάλιστα και οι προηγούμενε και όλοι οι αναφέρθηκαν σε πολύ σημαντικά ζητήματα που ελπίζω τελικά να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Είμαι σίγουρος ότι ο εισηγητής θα συμπεριλάβει τις περισσότερες προτάσεις των σχεδόν εισηγητών και θα υπερψηφιστούν από τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο αφορά το στόχο της έκθεσής μας. Ο ισχύων στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ποσοστά που έχει τώρα δεν αρκούν για να συγκρατήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 2 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το όριο των 2 βαθμών Κελσίου και να μην το υπερβούμε στην θέρμανση του πλανήτη, θέλουμε συμφωνίες εκπομπών στο Παρίσι πιο φιλόδοξες και από αυτές των εθνικών συνεισφορών ε, όπως έχουν δημοσιευθεί των INDCs. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους ε, στην, στη Σύνοδο των Παρισίων να είναι πιο φιλόδοξοι. Επίσης θα πρέπει να γίνει έγκαιρος η απαλλαγή μας από τις α, ε, ενώσεις και εκπομπές του Άθρακα. Αναφέρονται ήδη στα ψηφίσματα της Λίμα και της Βαρσοβίας θα πρέπει να μειωθούν και να εξαφανιστούν σταδιακά οι επιδοτήσεις ε, για τα αρκτά καύσιμα, ώστε να έχουμε μετάβαση σε μια ε, οικονομία ελεύθερη από άθρακα. Όσο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τα δικαιώματα των γηγενών πληθυσμών, των αυτόχθονων, ε, οι τοπικών κοινοτήτων. Να αποφύγουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τις κλιματικές μας δράσεις ως πρόσχημα για απεικιοκρατικές ε, δραστηριότητες, νέο απεικιοκρατικές. Θέλουμε κάποια μέτρα για το κλίμα που θα λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των αυτόχθων πληθυσμών, την ισότητα των φύλων και το καθεξής. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν με βάση τις ε, τοπικές τους παραδόσεις ε, και το σεβασμό των αυτόχθονων πληθυσμών τους. Και ένα τρίτο τομέα που αναφέρθηκε ήδη από τον κύριο Γκερμπάντη αφορά το θέμα της χρηματοδότησης του κλίματος, των κλιματικών δράσεων. Αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο της συζήτησης στο Παρίσι. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πακέτο. Χρειαζόμαστε αξιόπιστο πακέτο και μέτρα για την περίοδο μέχρι και μετά το 2020. Θα πρέπει να στηρίξουμε δράσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες και επίσης η, χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Και τέλος, χθε είχαμε συζήτηση με τον κύριο Κανιέτα στην Επιτροπή και πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τον κύριο Γκερμπράντι ότι χρήματα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κλιματικές δράσεις. Υπάρχουν, αλλά δεν διατίθενται για κλιματικές δράσεις. Τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών και γενικώ τα έσοδα τέτοια, τέτοια από, το, το κλίμα θα πρέπει να αφιερώνονται αποκλειστικά και μόνο για κλιματικές δράσεις. Αλλιώς δεν θα έχουμε αξιόπιστη διαπραγματευτική θέση στο Παρίσι. Ευχαριστώ κύριο Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Συμφωνώ μαζί του όταν λέει ότι για αυτό το θέμα ε, ισχύει μια γενική ευμένη συμφωνία και αυτό είναι παρηγορητικό γιατί ο στόχος είναι τόσο σημαντικός, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες εν ώψη της διάσκεψης του Παρισιού και είναι καλό να υπάρχει, καλή, ε, να υπάρχει συνένεση ε, των στόχων και των ιδεών που θα πάμε στο Παρίσι. Ακριβώς κάποιες παρατηρήσεις που θέλαμε να κάνουμε και θα, στόχους που θέλαμε με τις τροπολογίες που υποβάλαμε. Το πρώτο σημείο ήδη αναφέρθηκε μόλις ε, από τον συνάδελφο των Πρασίνων, ότι δηλαδή η επιστήμη μας λέει ότι ακόμα κι αν ε, οι δεσμεύσεις και οι στόχοι η ε, φιλόδοξη που έχουμε εμεί αναλάβει ω Ευρώπη, αλλά είδαμε πως ευτυχώς και άλλες χώρε σημαντικέ όπως η Κίνα, η ΙΠΑ, ακόμα και αν οι δεσμεύσεις αυτές διατηρηθούν και θα είναι δύσκολο να τηρηθούν, αν και, αν δεν τηρηθούν, δεν θα τα καταφέρουμε να μείνουμε εντό της ε, των δύο βαθμών. Η προσπάθεια είναι τεράστια, αλλά δεν αρκεί. Ε, και όταν λέγατε ότι η Ευρώπη έχει αφήσει πίσω τους άλλους, θα πρέπει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε και άλλες χώρες, οι άλλες ήπειροι, να ακολουθήσουν το παράδειγμα γιατί ακριβώς η προσπάθεια πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη από αυτήν που ήδη έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Να προσθέσω κάτι στις τροπολογίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και είναι παράλληλο με αυτή την προβληματική είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το λάβουμε υπόψη γιατί η ρυθμή ανάπτυξης που προβλέπονται είναι φουτρομακτική. 11 δις ε, άνθρωποι το 2030. Ε, ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά αυτά τα στοιχεία τα... Δεν, βασίζω, δεν θα πρέπει μάλλον το μέλλον το σκεφτούμε με τον πληθυσμό που έχουμε σήμερα, αλλά με το μελλοντικό πληθυσμό. Τεράστια ζήτηση ενέργειας, αύξηση ζήτησης από πλευρά όλου αυτού του πληθυσμού. Αυτό συνδέεται και με τις κλιματικές μεταναστευτικέ ροές και εδώ θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να δεσμευτούμε όσον αφορά τα μέτρα τα μέτρα που θα λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης θα πρέπει να περιμένουμε από το Παρίσι και οικονομική δέσμευση, δηλαδή πόροι ε, κονδύλια που κυρίως θα προέρχονται από τις πλουσιότερες χώρες και τις πιο υπεύθυνες χώρες για τις εκπομπές προς τις υπόλοιπες χώρες που μας ζητούν να αναπτυχθούν και εμείς τους ζητούμε να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο, όταν εμείς μέχρι στιγμής δεν το κάναμε αυτό. Άρα ε, είναι σωστό να βοηθηθούν για την προσπάθεια την επιπλέον που πρέπει εκείνοι να καταβάλουν λόγω των παλιών μας ε, ε, εμάς συμπεριφορών. Άλλο στοιχείο είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ίσως όσον αφορά τι ανανεώσιμες ενέργειες κάπως να έχουμε σταθεί και να πιέσουμε στις, τεχνολογίε τεχνολογίες που υπάρχουν ήδη, που είναι Πολλαπλέ και που δεν είναι αρκετά διαδεδομένε, αλλά γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν χώρε τη Μέση Ανατολή που αυτή τη στιγμή είναι, τεράστι... είναι μεγάλη εξαγωγή πετρελαίου και μα λένε ότι σε 20-50 χρόνια όταν δεν θα έχουμε πια πετρέλαιο να εξάγουμε δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί θα εξάγουμε ανανεώσιμε τεχνολογίε. Αυτοί δουλεύουν γι' αυτό με πολύ έντονου ρυθμού και η Ευρώπη θα μπορούσε να επενδύσει σε έρευνα και καινοτομία για να έχει και η ίδια, ε, να βρεθεί η ίδια στην πρωτοπορία για τι ανανεώσιμε. Για το ETS εμεί προτείναμε και για το θέμα επίση τη Ενεργειακή Ένωση, προτείναμε τουλάχιστον την ιδέα όχι μόνο να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να το αλλάξουμε, γιατί το ETS δεν έχει λειτουργήσει, δεν μείωσε τις εκπομπές και δεν βελτίωσε την ενεργειακή επάρκεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μελετήσουμε ένα εναλλακτικό σύστημα, γιατί αυτό δεν λειτουργεί. Δεν σημαίνει και ότι αν το τροποποιήσουμε θα λειτουργήσει. Ε, μάλλον χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό. Και τέλος, πέρα από τον ορισμό χρονικών στόχων που υπάρχουν, και εδώ εντάξει έχουμε κάποιες διαφορές απόψεων, Πάντως θα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει ε, να ζητήσει και ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσει για την επιτυχία αυτών των χρονικών στόχων και να κάνει και μια επαλήθευση από καιρού εις για να βλέπει αν προχωράμε στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς και εγώ χαιρετίζω το έργο του εισηγητή είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί ήδη. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε αυτά τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά που ελέγχα. Νομίζω ότι η COP21 θα πρέπει πράγματι να δώσει συγκεκριμένη υποστήριξη στις νέες τεχνολογίες με χαμηλή χρήση άνθρακος, να εντοπίσει ποιες είναι αυτές τις τεχνολογίες και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την ε, θέση σε λειτουργία των τεχνολογιών εδώ. Επομένως, θα πρέπει να παίξουμε και εμείς ένα σημαντικό ρόλο για την πρόθεση αυτών των τεχνολογιών και να τις λάβουμε υπόψη στα πλαίσια της COP21. Έχω προτείνει μερικές τροπολογίες ε, προς την κατεύθυνση αυτή, μαζί με κάποιους συναδέλφους μου, για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών διοξίδου του άνθρακος με την κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να βρίσκονται μέσα σε ένα κατάλογο προτινομένων λύσεων. Κάνει πολλές προσπάθειες η Ευρώπη στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει όμως να παραμείνουμε στα επίπεδα του πραγματιστικού ρεαλισμού. Έχουμε καθορίσει ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο του στόχους μας για το 2030. Κάποιοι θέλουν να προχωρήσουν εκεί ακόμα επέκεινα, 50% μείωση εκπομπών παραγωγής αλλά για το 2030 νομίζω πρέπει να παραμείνουμε σε επίπεδο ορατότητα σκεφτόμενοι και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να φέρουν σε πέρα σε αυτούς τους στόχους. Για μένα ο καλύτερος στόχος να πετύχουμε στο Παρίσι είναι να είμαστε φιλόδοξοι, όλοι το θέλουμε, αλλά και πραγματιστές. Και επιμένω σε αυτό το σημείο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με είχατε ξεχάσει, αλλά εγώ σας συγχωρώ. Κύριε ε, εισηγητά, σας ευχαριστώ για την έκθεση και τη στράτευσή σας στο θέμα αυτό που είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, του αιώνα ε, μας όπως μας υπερθύμισε και ο Πάπας. Αφορά τις, ε, τον τρόπο ζωή μας και τη σχέση μας με τη φύση. Το σχέδιο έκθεσης για το COP21 στο Παρίσι Ελπίζουμε να μην είναι απλώ ε, ένα επικοινωνιακό εγχείρημα και αυτό φοβάμαι και το λέω με κάθε σεβασμό προς το έργο σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά φαίνεται ότι πάμε προς ολοταχώ προς μια αποτυχία αντίστοιχη με τις ε, Κοπεχάγη το 2009. Ποιο θα ε, συσπηρωθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσπάθειε τη για τη μείωση των εκπομπών θα ξεχάσαμε τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Μην με παρεξηγείτε. Δεν θέλω να επιβάλλω συμφωνίε σε άλλε περιοχέ του κόσμου και σε άλλε χώρε για να εκβιάσω του πολέμου τη συμφωνία. Αλλά ούτω ή άλλω δεν έχουμε και τα μέσα για κάτι τέτοιο. Αλλά α το ομολογήσουμε. Και γι' αυτό υπέβαλα και σχετικέ τροπολογίε. Έχουμε το οικονομικό πλαίσιο και την πολιτική βούληση στην οποία στηρίζουμε τον αγώνα μα για το κλίμα. Αφενό, θα πρέπει να αποδεχτούμε την αποτυχία του υφισταμένου συστήματο, τουλάχιστον να ομολογήσουμε την ανεπάρκειά του. Γιατί? Γιατί απλούστατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε αισθητά τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου ε, και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, θα εκπέμψουν πολύ σύντομα πολύ περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από εμά. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα προβλήματα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μειωθούν οι εκπομπές τους ε, με αντίστοιχη μείωση της ε, ανάπτυξης τους, όπως συμβαίνει με εμά. Ούτε είναι έτοιμες οι χώρες αυτές να καθοτήσουν συστήματα ρύθμισης της ρήπανσης όπως κάνουμε εμείς, ε, γιατί προτιμούν να βλάπτονται μερικοί από ότι να ορίσουν ανώτατα όρια αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε όσο βλέπουμε το οικονομικό σύστημα υπό τη σκοπιά του παγκόσμιου γιγαντισμού, τόσο δημιουργούμε με κινδύνους παγκοσμίω. Δεν χρειαζόμαστε παγκόσμια ρύθμιση και μέτρα, αλλά πιο ε, περιφερειακές και τοπικές ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά την εγκύκλιο του ΠΑΠΑ, ε, αναφέρεται, αναφέρεται στην ιδεολογική έκθεση για την ηθική και πνευματική κλίση της Ευρώπης. Ελπίζω το ΕΛΚΑ αντίστοιχε θέσει να υιοθετήσει και για τα θέματα τη ζωή, τη οικογένεια ή απέναντι στο κοινωνικό δόγμα τη Εκκλησία. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Miss Ευχαριστώ κυρία Ντάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζιλ Παρνιό για την έκθεσή του που επικεντρώνεται σε πολύ σημαντικά θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αν θέλουμε να έλθει σε αίσιο πέρας COP21. Συμφωνώ ότι με την έκθεση αυτή έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά. Θα πρέπει βέβαια να διαπραγματευτούμε κάποιες συμφωνίες τριασμού των κλιματικών αλλαγών και να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να έχουμε όλο και λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο μέλλον. Κατέθεσα και εγώ κάποιες τροπολογίες. Οι μεταφορές είναι ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας που συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολιτικές για να μειώσουμε τις εκπομπές καυσαερίων από τις μεταφορές. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στις πιέσεις που θα πρέπει να ασκήσουμε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στην Διεθνή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ε, γιατί πολλές χώρες ε, βάζουν ένα τίμημα στην ρήπαση. Ο όπως με το σύστημα εμπορίας εκπομπών που έχουμε στην Ευρώπη ή αντίστοιχα συστήματα, θα θέλαμε ένα παγκόσμιο σύστημα. Γιατί αν συνεργαστούμε θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα είναι και πιο μεγάλες οι φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Επίσης θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα για τα τρόφιμα, το είδωρ και το έδαφος. Και ίσως το κλίμα αποτελέσει αιτία μαζικών μετακινήσεων στο μέλος. Κάτι που θα είναι πολύ αρνητικό. Γιατί με το κλίμα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και μάλιστα αηφόρο. Το γνωρίζει αυτό ο συνάδελφος. Ε, και θεωρώ ότι πολλές φορές κλίμα και μετανάστευση ε, είναι αλληλένδετες έννοιες. Γι' αυτό θα πρέπει το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε στην ρίζα του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να θετηθούν κάποιες δράσεις για να μετριαστεί η εκπομπή αερίων από τις θαλάσσιες μεταφορές για να βελτιώσουμε και το θαλάσσιο περιβάλλον και να μειώσουμε τη ρήπαση των θαλασσών. Έτσι θα επηρεάσουμε θετικά το περιβάλλον παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ο Ιβο Μπέλετ. Thanks very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά από τα οποία ελέγξαν. Και ο κύριος Πανιώτα έχει αναφέρει στην Επιτροπή Μεταφορών όπου ήμουν σκιώδης συγητής δύο παρατηρήσεις Καταρχήν αυτά που είπε ο κ. Φλόρας για ένα από του πιο πεπειραμένου βουλευτέ μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τι για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε στο Παρίσι με ευρία υποστήριξη από τις κύριε πολιτικές ομάδες. Όχι μονάχα μια πλειοψηφία για την έκθεση Παρνιό, αλλά να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και να πάμε στο Παρίσι ενωμένοι με μία μοναχαφωνή και να αποφύγουμε την πολυφωνία. Δεν είναι απαραίτητο. Πάντα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε υπερφιλόδοξοι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να περάσουμε τους στόχους για το 2030. Αν όμως βάλουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε ενωμένοι στο Παρίσι. Αυτό θα καλή ιδέα. Και επίσης από την Επιτροπή Μεταφορών, όπως το είπαν ορισμένοι συνάδελφοι και το είπε και η κυρία είναι σημαντικές προσπάθειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από τον τομέα της ναυτιλίας και, της, ε, και τον αεροπορικό κλάδο. Θέλουμε να ζητήσουμε να λάβετε υπόψη και τις προτάσεις της Επιτροπής Μεταφορών Έχουμε αναπτύξει κάπως περισσότερο την παράγραφο 10. Νομίζω ότι αυτές είναι καλές προτάσεις από την Επιτροπή Μεταφορών και να αναπτύξει υπόψη και τις περαιτέρω προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν από τον τομέα από τομείς πέραν των μεταφορών για καλύτερη ηλεκτροδότηση και καλύτερη ε, αποθήκευση της ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ευχαριστώ για το γεγονό ότι εξαίρεση και την ε, ε πείρα του Καλ Χάιντς Φλόρνς. Ο κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω δει λιγότερες προεδρίες από τον Καλ Χάιντς Φλόρενς, αλλά αυτό είναι και αυτό ένα επίτευγμα. Να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Ιβο Μπέλλες, γιατί μίλησε για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών γιατί εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά τα οποία λέει. Είναι μια καλή γνωμοδότηση με πολύ καλά σχόλια, ιδίω σε ό,τι αφορά τα θέματα του αεροπορικού και του ναυτιλιακού κλάδου, που ελπίζω ότι ο κ. Πάρνιο θα τα λάβει υπόψη. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η εκθέση, η οποία είναι πολύ καλή. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλα αυτά. Μόνο δύο <clears throat> ή τρει παρατηρήσει που θέλω να προσθέσω. Κάνει μια έκκληση το ΕΛΚ ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι με όλες τις πολιτικές ομάδες και βέβαια μετά προσπαθεί να περάσει τη δική του θέση σαν θέση ενωτική. Και εγώ στη θέση σας αυτό θα έκανα βέβαια. <clears throat> σας συγχαίρω λοιπόν για την πολιτική αυτή τακτική. Πρέπει να πω όμως ότι οι τωρινοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στην ομοφωνία στο Συμβούλιο. Έχουμε 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμφωνούν. Αν λέει το Κοινοβούλιο ότι αυτή είναι μια ενωμένη θέση μας δεν νομίζω ότι πράγματι ανταρακτούμε τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ας σταματήσουμε να είμαστε απλώς μια ακόμα περαιτέρω γραμματεία του Συμβουλίου. Ξέρουμε για την, από τις προτάσεις για το ETS ότι η Κομισιόν είναι απλώς η γραμματεία του Συμβουλίου. Ας μην παίξει λοιπόν και το Κοινοβούλιο τον ίδιο ρόλο μιας απλής γραμματείας. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποιες καλύτερες λύσεις. Και για τον κύριο Χέρμπραντ, ο οποίος έφυγε δυστυχώς, λέω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους στόχους μέχρι το 2020. Δεν ξέρω από πού έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τώρα το μείον 27% μειώσεων σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μέχρι το 2020. Ξεπερνάμε κατά πολύ τους στόχους μας. <clears throat> Δεν είναι λοιπόν αξιόπιστη η θέση μας για το Παρίσι και γι' αυτό έχουμε αυτό το τεράστιο αριθμό πιστοποιητικών για το σύστημα ETS και λέει η Κομισιόν πρέπει να πάρουμε από αυτά, αυτά τα πιστοποιητικά να περάσουμε από τη φάση 3 στη φάση 4 ώστε οι επιτυχίες μας που έχουμε για μειώσεις μέχρι το 2020 θα χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν την περαιτέρω πρόοδο μετά από το 2020. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν το Κοινοβούλιο να έχει μια πιο <clears throat> κριτική στάση και συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να δείξουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι καταλαβαίνουν καλύτερα τους αριθμούς και λένε γι' αυτό ότι θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο περισσότερη φιλοδοξία στους στόχους μας και σύμφωνα με το ΕΛΚ ότι θα έπρεπε όλοι να ενωθούν γύρω από αυτόν τον καινούριο πιο φιλόδοξο στόχο. καλό λοιπόν το ΕΛΚ να έρθει και αυτό στη δική μας πλευρά γιατί έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη προσέγγιση απόψεων όταν υπάρχει και και κίνηση από τις δύο πλευρές και προσβλέπω στον άρθει ο Καλ Χάντς προς τη δική μας άποψη με όλη την εμπειρία του. Τέλος για τη χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο είναι κέριο είναι να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για το τι προτείνουμε για τη χρηματοδότηση. Κάθε φορά που το λέμε αυτό, όταν τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, ας πούμε κάτι στις προτάσεις μας, ας πάρουμε τα έσοδα του ETS για να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή και όταν κάνει κάτι, γίνει κάτι για τον ε, τομέα της ναυτιλίας και της αεροπορίας, αυτά τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την ε, χρηματοδότηση του Ταμείου Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να έχουμε προβλέψιμους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε μια αξιόπιστη λύση στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Σούιτσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Παρνιέ, για την πολύ καλή του έκθεση. Εγώ είμαι ε, η, η συγκεκριά γνωμοδότησης της ΑΦΕΡ για το θέμα αυτό. Ε, χθε καταλήξαμε σε κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε, θα τι λάβετε σήμερα. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε πολύ καλέ συμβαστικέ λύσει. Σα ευχαριστώ πάντω για το νέο κεφάλαιο που προσθέσατε και που αναφέρεται στην κλιματική διπλωματία. Πολύ σημαντικό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Ελπίζω να λάβετε υπόψη, κύριε Παρνιό, και τι δικέ μα προτάσει σχετικά. Επίση, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το τονίζουμε αυτό ε, πολύ συχνά αναφέρονται αναφέρθηκα ε, τα λόγια του Πάπα, της Άγγελας Μέρκελ, όλα αυτά εμπίπτουν στην ευρύτερη έννοια της ε, κλιματικής διπλωματίας και χαίρομαι που υπάρχει σχετικό δάφιο σχετικά. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι θα πρέπει να μείνουμε συσπηρωμένοι, συμπαγείς, ενωμένοι στο Παρίσι και ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Γιατί θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και ταυτόχρονα να έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ελπίζω να συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο τάσεις για να συνεχίσει η Ευρώπη να λειτουργεί. Δεν είμαι κατά των στόχων, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που δεν άκουσα μέχρι στιγμής. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο TTIP Ξέρω ότι η Διατλαντική Συμφωνία δεν είναι το αντικείμενο αυτής της έκθεσης, αλλά μέχρι το 2015 θα έχουμε ήδη ε, καταλάβει το πνεύμα των διαπραγματεύσεων στο TTIP. Ε, ίσως λοιπόν ε, δεν θα πρέπει να ε, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτά που ήδη ακούγονται για το TTIP μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή. Ας το σκεφτεί ο εισηγητής. Επίσης, όταν μιλούμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, μερικές φορές ε, ελαφρά την καρδία μιλούμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, αλλά συμπεριλαμβάνουμε και αυτές και πλούσιες χώρες, όπως τη Σαουδική Αραβία, που δεν είναι καθόλου φτωχή. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε ίσως την ορολογία μας όταν μιλούμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάντως, ε, συμφωνώ ότι τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών να αφιερωθούν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γουέρφρεμ, για να μας πει τη γνώμη του για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τα σχόλιά μας. Γενικώ ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια θετική ε, στάση και δημιουργήθηκε και μία όθηση θετική για εν ώψη της COP21 και μάλιστα στις 29 Ιουνίου είχαμε και τις δηλώσεις της Κίνας για την COP21 και σήμερα περιμένουμε αίσια έκβαση της διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Και έχουμε και άλλες θετικές εξελίξεις ε, στο δρόμο προς το Παρίσι. Και πιστεύω ότι και οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμβάλλουν στο να γίνει έκθεση ένα ακόμη θετικό στοιχείο στη δημιουργία θετικού κλίματος και θετική όθησης εν ώψη των Παρισίων. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκάθαρη στάση και αυτό θα επιτρέψει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφανθεί με ενιαία φωνή. Διαπιστώνουμε αρκετά σημεία σύγκληση ε, στην έκθεση για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε την ανάγκη της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Θα πρέπει αυτά οι δύο να χαρακτηρίζουν τη Συμφωνία των Παρισίων, που είναι ε, κλειδιά για την αξιοπιστία με συμφωνίες ε, και δεν έχουν ε, ίσως αναφερθεί ιδεόντως, έχουν κάπως υποτιμηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. δεν νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ο κατάλληλο τόπο για να αμφισβητηθούν οι συμφωνίε μα για του στόχου μέχρι το 2030 και μετά. Αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε μεταξύ μα. Εν ευθέτω χρόνο, γιατί αφορούν εσωτερικέ μα πολιτικέ. Πάντως ε, θα έχουμε και επαφές με τους διεθνείς μας εταίρους και πριν και μετά το, και στο Παρίσι για τους στόχους μας και τα μέχρι τώρα επιτέγματά μας. Ακόμη και σε ό,τι αφορά το φόρουμ INDC για τις εθνικές ε, προκαθορισμένες συνεισφορές που θα ε, γίνει με συνδιοργάνωση της κυβέρνησης του Μαρόκου τον Οκτώβριο. Σίγουρα ε, η έκθεση είναι υποχρεωτικά σύντομη, γι' αυτό και χρειάστηκε να υποβληθούν τροπολογίε για να την εμπλουτίσουν. Χαίρομαι για τα, για συμπεράσματα του G7, για την καταπολέμηση της αποψήλωσης, ε, για την αναφορά της διπλωματίας για το κλίμα και για τον περιορισμό των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και αξιοπιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι και η χρηματοδότηση του κλίματος από τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό ε, ανήκει στην ε, βασική προσέγγιση μας. Είναι σημαντικό τη στοιχείο γιατί θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση του κλίματος συνδέεται άρρηκτα με την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επίσης ε, θέλουμε να δοθεί περισσότερο βάρος στη χρηματοδότηση της προσαρμογής και να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γιατί έχουν και αυτές επενδύσεις και ε, καινοτόμα αναπτυξιακά εργαλεία για να προσελκυστούν και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη και είδαμε κάποια θετικά μηνύματα για την διεύρυνση της βάσης των δωρητών. Βλέπουμε όλο και περισσότερες χώρες ε, του Νότου και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, να ε, έχουν κάνει κάποιες συμβολικές συνεισφορές στο Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο. Είναι πολύ θετική λοιπόν αυτή η συνεισφορά, όσο και είναι μικρή και συμβολική. Σας ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τη δευτερολογία του εισηγητή μας, του κυρίου Παρνιό. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, καθώς και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν τόσο αξιαγάπητος ε, και ευγενικό απέναντι στην έκθεση που μου συνέταξα. Πρόκειται για καλή βάση, είπατε όλοι, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω πως υπάρχει ανάγκη να βρούμε ε, κάποιες συμβιβαστικές, κυρίως όσον αφορά τους στόχους, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να είμαστε αξιόπιστοι, αλλά και να να είμαστε ε, αμόφωνοι. Και πέρα από αυτή την αξιοπιστία να μπορέσουμε να δώσουμε ως σύνολο, Συμβούλιο, Κομισιόν και εμείς στο Κοινοβούλιο, να μιλήσουμε με μια φωνή σε αυτή την ε, κόπ του Δεκεμβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ισορροπημένοι αλλά και ομοιογενείς για να είμαστε ισχυρότεροι ε, και αυτό είναι και το νόημα κάποιων συμβιβαστικών που θα δουλέψουμε όλοι μαζί στο πλαίσιο των επομένων συνεδριάσεων. και Επίσης, οι συγητές που εργάζονται για τη γνωμοδοτήση στην Ήτρε, στην Τραν, στην ΤΕΒΕ και στην ΑΦΕΤ, ο καθένας δηλαδή από τους εισηγητές για γνωμοδότηση, θα συμβάλλουν και θα πληθούν να συμμετέχουν στις 9 Σεπτεμβρίου στην επόμενη συνεδρίαση και έπειτα στις 14 Σεπτεμβρίου για την τρίτη συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές για να πάω και πιο γρήγορα. Τα θέματα που αντιμετωπίσαμε λοιπόν σε αυτές τις συνεδριάσεις ε, μας οδηγούσε περίπου 12 με 15 τροπολογίες συμβιβασμού να χαιρετήσουμε την ε, δήλωση των G7 και G8 για την αποανθρακοποίηση, την απανθράκωση της οικονομία. Δεύτερον, η πρόταση που αναμένεται στον αγώνα για την κατά της κλιματικής αλλαγής. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των επιστημονικών εμπειρογνωμοσυνών και της εφαρμογής, η δέσμευση των κρατών μελών για τη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλου του Κιώτου, ο κανονισμός σε σχέση με τις εκπομπές από τον αεροπορικό και ναυτιλιακό κλάδος, και η χρήση των εσόδων από αυτό το μέτρο, η χρήση του Πρασίνου Ταμείου, η βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων και τη συμμετοχή των τρίτων χωρών. Όλα αυτά είναι οι προοπτικές λοιπόν για την COP21. Από τις 230 λοιπόν αυτές τις τροπολογίες μπορούμε να καταλήξουμε σε μια σειρά τροπολογιών συμβασμού που πολύ εύκολα θα μπορέσουν να υποστηριχθούν και μετά έχουμε μια δεύτερη σειρά από συμβαστικές λύσεις. Είναι πρώτα απ' όλα ο καθορισμός στόχων για τη μείωση των παγκοσμίων εκπομπών <clears throat> αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το, αερίου θερμοκηπίου μέχρι το 2050 καθορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων για τη μείωση των εκπομπών μεταξύ 2.30-2.50 επανεξέταση της διαδικασίας μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κάθε πέντε χρόνια, καθορισμός περίοδων μείωσης από το 2050 και πέκυνα, προετοιμασία ενός χρηματοδοτικού πακέτου και η ανάγκη να προβλέψουμε καινοτόμε μορφέ χρηματοδότηση να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Άκουσα αυτά που είπε ο Καρλ Άιντ Φλόρεντ, και έχουμε πράγματι ένα κοινό στόχο να δημιουργήσουμε ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αλλά και πάλι θα είναι μια πρόταση η οποία δεν συλλέγει την ομοφωνία όλων και σήμερα όπως είπε ο Καλ Χάρνς μπορεί να είναι ένα εμπόδιο σε περαιτέρω συμφωνία γι' αυτό θα εξετάσουμε τις σχετικές τροπολογίες κάποιες μιλάνε για πρωτοβουλίες κάποιες Κάποιοι μιλάνε για ένα φόρο στα καύσιμα. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν υποφελώς για όλα αυτά τα θέματα στις διάφορες συνεδριάσεις μεταξύ εισηγητών και σκιωδών εισηγητών και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επιτρέψουμε να διατυπωθούν προτάσεις χρηματοδότησης οι οποίες θα είναι καινοτόμες και οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν τα δημόσια χρήματα να είναι στο ραντεβουδάκι. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι μπορούμε να προτείνουμε και τροπολογίες που αποτελούν πρόπτικες που επιτρέπουν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες μιας χρηματοδότησης ενώ εγγραφώνται σε ένα τοπίο χωρίς εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των βιομηχανιών που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και είναι φορείς ε, ελπίδος για το επόμενο επερχόμενο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω υπό μορφή συμπερασμάτων. Ευχαριστούμε πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. 22 <clears throat> Σεπτεμβρίου θα εγκρίνουμε στην Επιτροπή μας αυτή την έκθεση και στην Ολομέλεια μάλλον στις 14 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε άλλα σημεία στη μέση διάταξή μας. Σας εύχομαι καλές καλοκαιρινές διακοπές σε όλα τα μέλη της Επιτροπές και καλή ώρα αν προλάβετε βέβαια.